Buongiorno a tutti. Καλημέρα σε όλους. Πρωτού ξεκινήσουμε τις εργασίες μας για την πρωινή μας συνεδρίαση, θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσει προς τα μέλη της Επιτροπής μας. Πρώτον, κοινή συνεδρίαση η οποία θα λάβει χώρα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 26 Σεπτεμβρίου από τις 3 ως τις 6.30 προκειμένου να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την έκθεση ένα πλαίσιο πολιτικών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι αφού λάβαμε τις κατεξοδότηση πράξεις για το GMES, για τις οποίες 7 μέλη αντιτάχθηκαν, σύμφωνα με τους εσωτερικούς μας κανόνες θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και η ψηφοφορία αυτή θα λάβει χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2013. Προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών είναι η Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ας ξεκινήσουμε τώρα τις εργασίες μας όσον αφορά την σημερινή δημόσια ακρόαση. Ξεκινήσαμε με μια μικρή καθυστέρηση γιατί ε, περίμενα να φτάσουν ορισμένοι συνάδελφοι. Ξέρετε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δημόσια ακρόαση στις 11. Ας προσέχουμε λοιπόν λίγο τον χρόνο, τον χρόνο ομιλίας. Η σημερινή δημόσια ακρόαση διοργανώθηκε από την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Βιομηχανίας και θα ασχοληθεί με ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω για τη βιομηχανική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι στη διαστημική πολιτική. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και αυτό είναι ο βασικός κινητήρας που έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει περισσότερο τον τομέα αυτό, στον οποίο έχουν ε, καταβληθεί πολύ σημαντικές προσπάθειες, ιδίως στο διακυβερνητικό πλαίσιο, στα πλαίσια της ΕΖΑ δηλαδή, και σε εθνικό επίπεδο με τις εθνικές υπηρεσίες διαστήματος. Την τελευταία δεκαετία καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ισχυρή βιομηχανική πλέον βάση και μπορούμε πλέον να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να δημιουργεί κάποιες διαστημικές τεχνολογίες, κάποιες διαστημικές εφαρμογές, ακόμα και τις δικές της πλατφόρμες εκτόξευσης. Υποστηρίζουμε λοιπόν εμείς την διαστημική αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των δύο βασικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοπέρνικους και τον Γαλιλαίο. Η σημερινή δημόσια ακρόαση θα στο Γαλιλαίο και τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα όσον αφορά τον κανονισμό του Γαλιλαίου. Ο κύριος Μαρινέσκου είναι συγητής ε, για τον κανονισμό αυτό. Μάλιστα πετύχαμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και νομίζω ότι μείναμε όλοι ικανοποιημένοι. Η ψηφοφορία στην Ήτρε θα γίνει την επόμενη μάλιστα εβδομάδα. Η διαστημική βιομηχανία μπορεί ε, πραγματικά να καταφέρει να υποφεληθεί πάρα πολύ από τον Γαλιλαίο και μπορούμε να έχουμε ωφέλη σε όλη την ε, βιομηχανική αλυσίδα. Πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί να γίνει μέσω του διαστημικού επίσης τομέα. Όπως λέγεται στην έκθεση της κυρίας Νίμπλερ, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανία δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό ποσό κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και απασχολεί περίπου 34.000 ανθρώπου. Το Γαλιλαίο και το Έγνος έχουν μεταξύ τους ένα πολύ αποτελεσματικό συντονισμό και οι πρώτες λειτουργίες του Γαλιλαίου θα εμφανιστούν πάρα πολύ σύντομα. Θα αρχίσει πολύ σύντομα να λειτουργεί πλήρως το σύστημα Γαλιλαίου. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά με τον οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS, GSA και ακόμη συγγήτρια για τον κανονισμό GSA, όπου προσπαθούμε μέσω του κανονισμού αυτού να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ε, οργανισμού GSA όσον αφορά την πιστοποίηση και την ασφάλεια. Είμαι στη διάθεσή σας για να δεχθώ και τις τροπολογίες σας. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αύριο 19 Σεπτεμβρίου είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών. Η συνάδελφος Νίμπλερ είναι υπεύθυνη για μία έκθεση πρωτοβουλίας η οποία ασχολείται με τα ωφέλη τα οποία η διαστημική βιομηχανία μπορεί να αποφέρει για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν άμεσα τη σημερινή μας συνεδρίαση. Έχουμε δύο πάνελ, δύο βασικά θέματα συζήτησης και θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στην συνάδελφό μας, την κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Δεσδορίδες, κύριε Ρόλφ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, και από τη δική μου την πλευρά να σας καλημερίσω Χαίρομαι που θα συζητήσουμε σήμερα ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που μπορέσαμε να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Σαρτόρη, που μας βοήθησε σε αυτό. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο παρελθόν πάντα ζητούσαμε μια πολιτική φιλόδοξη για το διάστημα. Θυμάμαι πάρα πολλά ψηφίσματα, πάρα πολλές αποφάσεις, εκθέσεις που συντάξαμε για να τονίσουμε πόσο σημαντικό θεωρούμε να υπάρχει μια ε, διαστημική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα τμήμα αυτής της φιλόδοξης πολιτικής είναι και το ε, κεφάλαιο που αφορά στην διαστημική βιομηχανία. Ο ε, Επίτροπος Σταγιάννη που θα έρθει αργότερα εδώ θα μιλήσει και για το θέμα αυτό γιατί η Κομισιόν νομίζω ότι επεξεργάζεται ακριβώς αυτό το θέμα πώς μπορούμε από τον Καλλιλέο και τον Κοπέρνικο να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε εντατικά αυτό το θέμα. Για μένα είναι σημαντικό και θέλω να το πω από την αρχή της ακροασής μας ότι το Γαλιλαίο θα πρέπει να τεθεί σε, σε χρήση και βεβαίως θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το Κοπέρνικος. Είναι οι ναυαρχίδες της πολιτικής μας. Έχουμε ε, φιλόδοξους ε, στόχους. Ε, μπορούμε να, θα, πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε το Γαλιλαίο προς χρήση από το 2014. Παράλληλα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε το πρόγραμμα Γαλιλαίο, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, στους πολίτες, ε, ε, γιατί, τι σημαίνει το Γαλιλαίο, γιατί ζητούμε χρήματα από τα κρατημέλη για να εφαρμοστεί. Όλοι ξέρουν το σύστημα GPS των Αμερικανών. Ε, αν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα ή ετοιμότητα ή διαθεσιμότητα για να, για να εξευρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις, ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό εμείς. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε ποια είναι η σημασία αυτών των ε, επιτευμάτων στους πολίτες μας. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι ευρωπαϊκές υπηρεσίες και μπορούν να κινητοποιηθούν εδώ εντός της Ευρώπης. Επίσης, θα δούμε το θέμα της ε, εμπορικής σημασίας. Ποια είναι η συμβολή του Γαλιλαίου και οι υπηρεσία του Γαλιλαίου ε, στην ε, οικονομία και μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι, τι ρόλο μπορούν να παίξουν αυτές οι υπηρεσίες έτσι ώστε να βοηθήσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ καλούς ομιλητές για την ακρόασή μας. Καταρχάς στο πρώτο πάνελ θα μιλήσουμε για το διάστημα ως ε, μηχανή ανάπτυξης ε, της ε, οικονομίας και χαίρομαι που έχουμε τον εκτελεστικό διευθυντή της υπηρεσίας GSA, τον κύριο Ντεσδορίδας, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και θα συζητήσουμε μαζί του και επίσης να καλωσορίσω και τον κύριο Κλάους Herbert Rolf που είναι διαχειριστικός διευθυντής της Class Agro Systems. Θα μας δώσει λοιπόν την άποψη της βιομηχανίας για το ποια είναι η συμβολή που μπορεί να έχει η διαστημική βιομηχανία, η διαστημική πολιτική για την ανάπτυξη για την οικονομία στην Ευρώπη. Στο δεύτερο πάνελ, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα μιλήσουμε για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως ε, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τον Γαλιλαίο και τις υπηρεσίες που απορρέουν από αυτό. Γιατί ε, από εκεί ε, εκπίπτουν πάρα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να το συζητήσουμε, να το σκεφτούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε αν υπάρχει πολιτική αναγκαιότητα, να δούμε αν πρέπει να παρέμβουμε έτσι ώστε ε, το, τη διαχείριση των, ε, ε, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να μπορούμε και από πολιτική πλευρά να την προστατεύσουμε. Στο δεύτερο πάνελ λοιπόν θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα στο 2013, ακριβώς λίγο πριν αρχίσουν να προσφέρονται οι υπηρεσίες του Γαλιλαίου, μπορούμε να ασχοληθούμε με τόσο σημαντικά ζητήματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα περάσουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ώρες. Αυτά από μένα. Και να α, ρωτήσω την κυρία Πρόεδρο, ε, θέλετε να, σας δώσω κατευθείαν το λόγο, θέλετε να αφήσουμε τον κύριο Δεσδορίδες να μιλήσει. Νομίζω, να, καταρχάς να ευχαριστήσω και να αφήσω την Πρόεδρο να μιλήσει. Ε, Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ για την εισήγησή σας και θα ξεκινήσουμε αμέσως με το πρώτο πάνελ, το πρώτο σύνολο μιλητών που έχει ως θέμα τον χώρο ως κινητήρια για την οικονομία και την οικολογική ανάπτυξη ε, και δίνουμε τον λόγο στον κύριο Ντεσδορίδης. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριοι, κύριοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ε, είναι τιμή μου σήμερα να σας δώσω την οπτική της ε, υπηρεσίας ε, GSA για, καθώς και το τι σημαίνουν όλα αυτά για την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι ώστε να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία το διάστημα και η διαστημική τεχνολογία και οι εφαρμογές είναι τώρα στα χέρια της αγοράς και σχεδιάζονται τακτικά. Πριν από πέντε χρόνια ακόμα υπήρχαν αμφιβολίες για το κατά πόσο όλες αυτές οι τεχνολογίες θα έμπαιναν τόσο γρήγορα στην καθημερινή μας ζωή. Το GNSS έχει γίνει ένας ε, παγκόσμιος φορέας για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Δύο δις ε, ε, έξυπνα τηλέφωνα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται με δυνατότητες GNSS και αναμένεται ότι στα επόμενα 10 χρόνια η, το ποσοστό διείσδυσης του GNSS θα διπλασιαστεί από το 30% που είναι σήμερα στο 60% περίπου. Δύο στα τρία δηλαδή από τα κινητά τηλέφωνά μας θα ε, ε, ε, περιέχουν την δυνατότητα GNSS. Σήμερα το 1 τρίτο των αυτοκινήτων στην Ευρώπη είναι εξοπλισμένα με το GNSS και τέτοιου είδου συσκευέ. Οι δορυφόροι στηρίζουν τις προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορία στι πόλει και να ε, μολύνεται έτσι, ρηπαίνεται μάλλον και ε, ε, λιγότερο το περιβάλλον. Οι χρήσεις γίνονται στην ναυσιπλοεία, στην αεροπλοεία, στην, στους σιδηροδρόμους και οι επενδύσεις στα συστήματα πλοήγησης και στις υπηρεσίες πλοήγησης μεσοδορυφόρου έχουν ήδη επιφέρει και θα εφέρουν ακόμη πολλές απτές αλλαγές στην αγορά. Ας εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα νούμερα. Παρά το γεγονός ότι η οικονομία μάλλον παρά την οικονομική κρίση, το συνολικό, τα συνολικά έσοδα από την αγορά για το GNSS αναμένεται να αυξηθούν στα επόμενα χρόνια κατά μέσο όρο ανά 9% ετησίως. Η μεγαλύτερη αναμενόμενη μεγέθυνση θα είναι σε χώρου, σε, για τις υπηρεσίες ε, εντοπισμού τοποθεσίας καθώς και σε οδικές υπηρεσίες. Αυτά τα δύο μαζί θα αποτελούν πάνω από το 90% της αγοράς. Σύμφωνα με τον ε, ΟΣΑ, κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στο διάστημα αναμένεται να φέρει ε, τέσσερις με νέα φορές περισσότερα στην αγορά ευρώ. Μακροπρόθεσμα λοιπόν αναμένεται ότι η απόδοση μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη. Κάθε ένα ευρώ που επενδύουν οι δημόσιες αρχές στο GNSS με βάση το ε, FES σύστημα μεταφορών μπορεί να ε, έχει ως κέρδος σύμφωνα με τη δική μας ανάλυση 10 ευρώ για την οικονομία. Αυτό αποδεικνύει ότι το, περισσότερο, το μεγαλύτερο τμήμα ε, της αγοράς GNSS έγκυται στις παρεπόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, η εμπλοκή της βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι θέματα κλειδιά για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως ε, την υποδομή GNSS της Ευρώπης. Η απόδοση των επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη και τι οικονομικές και κοινωνικές ε, απολαβές, δηλαδή περισσότερη απασχόληση, μεγαλύτερη απόδοση για τις επιχειρήσεις, κόστος και ωφέλη. Ε, μέσα στα επόμενα 14 χρόνια τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη από την έγνωση και την Γαλιλαίο και τον Γαλιλαίο υπολογίζονται σε 9 δις ε, ευρώ. Πράγμα που συμπεριλαμβάνει και κέρδη όπως η μείωση του χρόνου ταξιδίου, η μείωση των εκπομπών ε, να ειρήνω από τα καύσιμα κτλ. Σήμερα χιλιάδες κόσμος εργάζονται στον τομέα ε, ε, του διαστήματος Εκτιμάται ότι περίπου το 50% των εργαζομένων στον τομέα ασχολούνται με το GNSS και τις ε, απορρέωσες θέσεις. Υπάρχει ζήτηση όχι μόνο για μηχανικούς και επιστήμονες, αλλά και για ειδικούς ε, της πληροφορικής, ε, ειδικούς στο business και όλες τις σχετικές ικανότητες. Αυτό σημαίνει πως η Ευρώπη γύρω από αυτά όλα οικοδομεί η Ευρώπη τεχνολογική τεχνογνωσία και βρίσκεται στο προσκήνιο των ε, βιομηχανικών ικανοτήτων. Είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε αυτό γιατί με το Γαλιλαίο η Ευρώπη επενδύει στις ε, τελευταίες ε, τεχνογνωσίες, τις πιο προηγμένες τεχνογνωσίες. Όλα αυτά στην αρχή ε, έχουν σχεδιαστεί για πολιτική χρήση και μπορούμε να αναμένουμε αυξανόμενη χρήση στην Ευρώπη χάρη στο ευρωπαϊκό GNSS. Ρόλο, ποιος είναι ο ρόλος τώρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας GNSS στην προώθηση της χρήσης του GNSS. Η υπηρεσία μας έχει εργάζεται μάλλον αόκνος για να επιταχύνει τη χρήση και να προωθήσει τη χρήση των ε, υπηρεσιών έγνωση και γαλιλαίο. Επίσης βασιζόμαστε σε ένα θετικό οικοσύστημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες ώστε να αποκομίσουν τα ωφέλη αυτών των δύο προγραμμάτων. Το εγγύς μέλλον περιλαμβάνει νέες προπτικές για την ανάπτυξη της αγοράς και ε, καταρχήν σημαίνει τη στήριξη της καινοτομίας μέσω του ορίζοντα 2020 και οικοδόμηση ισχυρού, ε, ισχυρής ε, εμπορικής τεχνογνωσίας. Δεύτερον, να αποκομίσουν ωφέλη όλοι ε, οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα μέχρι την υιοθέτηση του GNSS. Αυτό είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα της, της GNSA, δηλαδή διάλογος με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς και τρίτον ανάπτυξη το τμήματο των χρηστών ώστε να προετοιμαστεί η ευρύτερη υιοθέτηση του συστήματος GNSS να τονίσω κάποια αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής. Καταρχήν, μπορούμε να αναφερθούμε στην πολιτική αεροπορία. Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες ωφελούνται ήδη από την διαδικασία προσέγγισης με τα μέσα έγνος. Έχουμε σήμερα 87 αεροδρόμια στην Ευρώπη που ωφελούνται από το σύστημα έγνος που είναι το σύστημα πρόδρομος του Γαλιλαίου. Χάρη στην δράση της ανάπτυξης στην αγορά της CC και του GNSA, ε, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων γεωργών χρησιμοποιούν ήδη το GNSS στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε προσιτή ακρίβεια και το έγνος έχει συμβάλει στο να εκδημοκρατιστεί η γεωργία ακριβίας και να αυξηθεί η χρήση και στην Ανατολική Ευρώπη. Και αυτά όλα θα τα αναπτύξει σε λίγο και ο κύριος Ρόλφ Κλάους Χέρμπερ. Στην επόμενη δεκαετία το GNSS που χρησιμοποιείται στους σιδηροδρόμους θα χρησιμοποιείται ακόμη περισσότερο. Θα υπάρξει δηλαδή μεγάλη αύξηση και αναμένεται ότι το 30% των σειρμών θα είναι εξοπλισμένο πολύ σύντομα με συσκευές GNSS. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GNSA εργάζεται για την υιοθέτηση του GNSS και του EGNOS στις οδικές μεταφορές, σε κατασκευές στην ε, αυσιπλοεία και ούτω καθεξής. Έχουμε ήδη ένα σημαντικό αποτέλεσμα ότι περίπου δηλαδή 30% των ε, υφιστάμενων ε, μοντέλων δεκτών έχουν, έχουν υιοθετήσει τον του Είναι σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα δεδομένου του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η ανάπτυξη του συστήματος να τη υπογραμμίσω άλλη μία σημαντική παράμετρο που είναι οι ρυθμιστικές δράσεις. Είναι εξίσου σημαντικές ώστε να κινητοποιηθεί η βιομηχανία του GNSS να συμπεριλάβει τον Καλλιλέο και ιδιαίτερα για την ε, ευρύτερη μαζική αγορά. Ε, σημαντική αναφορά θα μπορούσε να γίνει στην, ε, στον κανονισμό e-call, όπου κάθε νέο είδος επιβατικού αυτοκινήτου και ελαφρού οχήματος θα πρέπει να έχει ένα σύστημα GNSS για ταχεία βοήθεια. Ε, σημαίνει αυτό ότι πάνω από 200 εκατομμύρια αυτοκίνητα καλύπτονται από αυτό τον κανονισμό. Ο κανονισμός ψηφιακού ταχυγράφου επίσης θα καλύψει πάνω από 30 εκατομμύρια φορτηγά που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή ε, στην Ευρώπη. Επίσης ο κανονισμός του 112 ε, για τις ε, πήγουσες καταστάσεις σημαίνει τον εξοπλισμό των εφιών κινητών τηλεφώνων με το σύστημα GNSS. Προσπαθούμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε και την αγορά, την υιοθέτηση μάλλον από την αγορά μέσω αριθμιστικών μέτρων. Τέλος να πω ότι το Γαλιλαίο εντάσσεται σε ένα πολύ ανταγωνιστικό σενάριο που άλλα συστήματα που υπάρχουν ή έρχονται και όπου η τεχνολογία χρήσης του εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ε, αναζητούμε εργαλεία και πόρους μέσω και πέρα από τα ερευνητικά μας προγράμματα για να στηρίξουμε καινοτόμες ιδέες στην Ευρώπη με υψηλό δυναμικό ε, εμπορίας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα να μοχλεύσουμε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως το ορίζοντας 2020 ώστε να οφείσουμε ε, επιχειρηματικές δράσεις δράσεις στην άκρη της αλυσίδας της αγοράς, ε, ώστε το Γαλιλαίο να φέρει ανταγωνιστικά πλονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα συστήματα. Είμαι πεπισμένος ότι με την χρήση του έγκνο και του Γαλιλαίου η ανάγκη για αριθμιστικές δράσεις και, και, και αντίστοιχοι πόροι για την ανάπτυξη των εφαρμογών GNSS βρισκόμαστε στο δρόμο ώστε να, ε, να μπορέσουμε να δράξουμε όλα τα ωφέλη που έχουμε προβλέψει για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ σα ευχαριστώ πολύ Κάρλο Ντορίδες για την εισήγηση αυτή και τώρα το λόγο θα πάρει ο Κλάου Έρμπερτ Ρόλφ που είναι Διευθυντής Μάρκετινγκ Asargo Systems. Ευχαριστώ. Χωρί μικρόφωνο μιλητή, όμω δεν τον ακούμε. Μικρόφωνο. Oh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέκα λεπτά μου είπατε. Ε, για αυτό το θέμα θα μπορούσα να μιλάω δύο ώρες βέβαια, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω μέσα σε δέκα λεπτά. Η γεωργία και η τεχνική των ε, ε, δορυφόρων ε, μάλλον δεν είναι κάτι καθημερινό για πολλούς από εσάς. Σε τέσσερα τμήματα θα ήθελα να χωρίσω τη δική μου παρουσίαση. Θα σας μιλήσω για τις τάσεις, μετά θα σας παρουσιάσω ποιοι είμαστε εμείς, η κλάς. Μετά θα μιλήσω γενικώ για την έξυπνη γεωργία, που πάντα όλο και περισσότερο τη βλέπουμε στις εφημερίδες και τα περιοδικά. Και μετά θα μιλήσω για το πού πάμε από εδώ και μπρος. Λοιπόν, τι μας κινεί. Έχουμε περίπου 7,1 δισεκατομμύρια άτομα ε, πληθυσμό στον ε, πλανήτη. Το 2050 θα φτάσουν τα 9 δισεκατομμύρια. Η ανάγκη λοιπόν για τρόφιμα και για κρέας αλλά και για σιτηρά θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Το ξέρουν οι πολίτες μας αυτό παγκοσμίω. Και βεβαίως ταυτόχρονα χάνουμε και επιφάνειες ε, αρρώσιμης γης που δεν μπορούμε να επαναφέρουμε. Έχουμε λοιπόν πολύ λιγότερες ε, γης για να ταΐσουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Εμείς ως κλάς κάνουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ε, παράγουμε διάφορα είδη αγροτικών μηχανών, ελκυστήρες, άλλες άλλου είδους μηχανές. Τα συνδυάζουμε και με τη σχετική τεχνολογία και πληροφορική ο καθηγητής ε, Ράντελ Μάχερ είχε αναφέρει ότι ε, πρέπει να ε, μπορούμε να ταΐσουμε τους πολίτες σε αυτού του κόσμου εάν χρησιμοποιήσουμε κάθε τετραγωνικό της γης πιο έξυπνα. Εδώ βλέπετε την έξυπνη γεωργία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εικόνα αυτή γιατί δείχνει πόσο, ψηφιακή έχει γίνει, πόσο ψηφιακός έχει γίνει ο κόσμος γύρω, γύρω μας. Τα πάντα είναι ψηφιακά πια σήμερα. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι δεν μπορούμε να γινόμαστε συνέχεια πιο μεγάλοι, πιο δυνατοί, δεν γίνεται να είμαστε όλο και πιο μεγάλοι όπως βλέπετε εδώ σε, κάποιες, σε αυτές τις εικόνες υπάρχουν και κάποια όρια πάντα στο πόσο μπορούμε να πάμε μακριά ε, πρέπει λοιπόν οι μηχανές μας να είναι πιο έξυπνες. Ο προηγούμενος ομιλητής ε, είπε ότι από το έγνος και το GNSS μέχρι τον Γαλιλαίο είναι ο σωστός δρόμος για να προχωρήσουμε. Ο Γαλιλαίο βέβαια είναι μόνο ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ο Κοπέρνικος, το οποίο θα ε, έρθω αργότερα. Αυτό το μοντέλο λοιπόν σας δείχνει και υποθέτω ότι το έχετε, το έχετε και τα έντυπα μου, μπορείτε να τα δείτε αν θέλετε. Βλέπετε λοιπόν εδώ ποιες είναι οι πιθανές μελλοντικέ τάσεις και οι τωρινές τάσεις που έχουν να κάνουν με ε, ε, τεχνολογία που βασίζεται στους δορυφόρους. Τώρα, από την πλευρά της γεωργίας, εγώ ως επιχειρηματίας θέλω να μπορώ να βλέπω από κάποιο συγκεκριμένο ύψος την, ε, ε την καλλιεργιά μου. Έχουμε ας πούμε μια καλλιέργεια στην Γερμανία ή, στην, ή σε κάποια άλλη χώρα. Και πολύ συχνά ε, έχουμε παραγωγή χείριου κρέατος ή παραγωγή γάλακτος, η οποία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 15% και θέλουμε να, το, ε, να, να έχουμε έναν έλεγχο όλη αυτή τη κατάσταση. Και αυτό θέλουμε να το πετύχουμε και μπορούμε. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε τους δορυφόρους, γι' αυτό χρειαζόμαστε πλοήγηση, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις συγκεκριμένε συσκευές και μηχανήματα. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε όμως να τον απελευθερώσουμε από πράγματα που είναι ανόητα. Να απελευθερώσουμε τον αγρότη από πράγματα που του δυσκολεύουν τη ζωή. Τον οδηγό τον, ε, της, ε, του μηχανήματος ε, τον χρειαζόμαστε γιατί ξέρει καλύτερα την τεχνολογία και μπορεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα να κάνει αυτό που παλαιότερα θα γινόταν πιο δύσκολα. Τώρα, η διαφάνεια. Οι πολίτες θέλουν όλο καλύτερη ε, χαρτογράφηση, όλο, καλύτερη, όλο καλύτερες πληροφορίες για τα τρόφιμα που χρησιμοποιούν και αυτό το νέο κοριτσάκι εδώ, αυτή η μικρούλα στην ε, φωτογραφία, θέλουμε με ασφάλεια να μπορεί να πίνει το γάλα της και να τρώει το ψωμί της και τώρα και στο μέλλον. Και αυτό που μπορούμε να για το μέλλον είναι αυτό που βλέπετε εδώ στην, ε, στη διαφάνεια. Δεξιά βλέπετε έναν δορυφόρο Γκαλιλαίο και στα αριστερά βλέπετε έναν ε, δορυφόρο του Κοπέρνικου. Ή τέλο πάντων όπω θα έχει ένα δορυφόρο του Κοπέρνικου. Και δύο πράγματα γίνονται για αυτό, το, για αυτό τον ελκυστήρα. Αριστερά δείχνει ποια είναι η εξέλιξη της βιομάζας στην καλλιέργεια. Οπότε με τους δορυφόρους μπορούμε κάθε έξι μέρες να έχουμε νέα δεδομένα για τη βιομάζα των φυτών. Μπορούμε πολύ νωρίς να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ζημιές λόγω παγετού, ενώ κανονικά χωρίς τους δορυφόρους δεν είναι εύκολο να το δούμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε λοιπόν με τις ε, τεχνολογίες αυτές να βελτιωθούμε. Δεύτερον, ο άλλος δορυφόρος, στα δεξιά όπως βλέπετε, δείχνει το δρόμο. Από το έγνος, ε, ε, μέσω του έγνος με πολύ συγκεκριμένη ακρίβεια και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή μέσα σε, μέχρι, μέχρι ακρίβεια 2 ε, εκατοστών. Υπάρχουν πολλά ε, ερωτήματα βεβαίως ε, για το τι χρειαζόμαστε την τόση ακρίβεια στην, στην Γεωργία. Πάντα στις, στη Γεωργία υπάρχουν, υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν χάρτες, δεν υπάρχει χαρτογράφηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ακριβεί στα δεδομένα που χρησιμοποιούμε. Και τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον. Όταν αν όλοι οι Ευρωπαίοι οι έχουν, μπορούν να βελτιώσουν αυτή την ακρίβεια κατά 5%, Σημαίνει ότι είναι σαν να μπορείτε να, να πετάξετε 23.000 φορές από το Παρίσι στο Βερολίνο. Μπορούμε δηλαδή να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ δυναμικό και αυτό είναι το καλό στο δικό μου το επάγγελμα. Μπορώ να βοηθήσω τους α, γεωργούς και μπορώ εγώ να πάω σπίτι μου ήσυχο το βράδυ και να πω στην κόρη μου σήμερα έκανα κάτι για το μέλλον σου. Έχουμε τα λοιπάσματα, έχουμε χημικά, χημικές ουσίες, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά από τη χρήση αυτών και αυτό είναι καλό. Και κλείνοντας, πολύ σύντομα να μιλήσω για το Κοπέρνικους και το σύστημα Κοπέρνικους, ε, τι ακριβώς μας περιμένει. Ε, δυστυχώς ε, υπήρξε μια καθυστέρηση τριών μηνών, η οποία τελικά κατέληξε να γίνει καθυστέρηση ενός χρόνου. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και μπρος. Έχουμε εταίρους που από το 2014 ήθελε να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα που είχε κατασκευάσει, δεν γίνεται να τα χρησιμοποιήσει επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η καθυστέρηση. Εν πάση αυτό είναι λίγο εκνευριστικό, αλλά ελπίζω ότι το 2015 θα καταφέρουμε να είμαστε λειτουργικοί ως προς τον Κοπέρνικους. Έχω κάποιες εικόνες εδώ να σας δείξω. Εδώ βλέπετε... Ε, η δεξιά εικόνα, όπως βλέπετε εσείς, είναι ε, ο δυναμικός χάρτης του AgroCom.net. Η μεσαία εικόνα είναι η εικόνα που βλέπετε από ραντάρ, έτσι όπως την παίρνει το ραντάρ. Δηλαδή αυτή την εικόνα θα δίνει ο Κοπέρνικος όταν θα είναι λειτουργικός. Και επίσης ε, μπορούμε να δούμε και τη διαφορά ή την ε, ε, ισοδυναμία των εικόνων. Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και από τον Κοπέρνικο και από τον Καλλιλέο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν η κυρία Νίμπλερ θέλει να πάρει το λόγο. Όχι, μάλιστα. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσα ακούσαμε πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Και είναι σαφές ότι επιθυμείτε να καταστήσετε όλες αυτές τις εφαρμογές πιο αποτελεσματικές. Αν όμως το σύστημα είναι άκαμπτο, δεν παρουσιάζει ευελιξία και δεν υπάρχει μια εναλλακτική λύση, τότε ένα άκαμπτο σύστημα είναι ένα σύστημα που όλα θα πρέπει αν υπάρχει έστω και ένας μικρός σύνδεσμος στην αλυσίδα που δεν λειτουργεί σωστά, τότε το όλο σύστημα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Και εγώ έχω εντοπίσει ή βλέπω τουλάχιστον δύο πιθανούς κινδύνους στο όλο σύστημα όπως το περιγράψατε. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε κακές καιρικές συνθήκες στο διάστημα. Ή ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα ηλιακά φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη σωστή λειτουργία των πραγμάτων στο διάστημα. Και στη συνέχεια υπάρχουν βέβαια και οι κίνδυνοι ανθρωπογενείς. Οι δορυφόροι σας ενδεχομένως να καταστραφούν εξαιτίας της σύγκρουσης του συντορυφόρου με κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία περιστρέφονται στο διάστημα. Στην περίπτωση αυτή καταλαβαίνετε ότι διηγούμεθα σε ένα πλήρες blackout. Τίποτα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπραζίτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω την ακόλουθη ερώτηση. Προέρχομαι από την Τσεχία και στην ε, δική μου τη χώρα και μάλιστα στις πιο έφορες περιοχές της χώρας μου χρησιμοποιούμε το σύστημα GPS για την εφή γεωργία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Για ποιο λόγο η δική σας προσφορά είναι καλύτερη, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δικού σας συστήματος σε σχέση με το σύστημα GPS. Η γεωργία ακριβίας η οποία θα βασίζεται σε ακριβείς εφαρμογές δορυφορικές, η οποία βασίζεται σε εικόνες GPS από δορυφόρους, είναι κάτι το οποίο ήδη το γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε στην Τσεχία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε, ξέρετε, στη χώρα μου πολύ μεγάλες γεωργικές εκτάσεις, και οι γεωργοί χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό το GPS. Με αυτό είναι εξοικειωμένοι. Για ποιο λόγο το δικό σας το σύστημα είναι καλύτερο. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, τότε να δώσω το λόγο στον κύριο Δεσδορίντες πρώτα για μια πρώτη απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, για, για το δεύτερο μάλλον ο κύριος Ρόλφ είναι καλύτερα εξειδικευμένος για να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά την, ε, ε, ε, αυτό το στεναρό σύστημα που έχουμε. Είναι καλό να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα του Γκαλιλαίου, γιατί ο Γκαλιλαίο μπορεί να συνδυάσει την απόδοση του υπάρχοντος συστήματος GPS θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να συμπληρώσει, να ενισχύσει το σύστημα του GPS. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που ήδη αναγνωρίζουν και οι συνάδελφοι από την άλλη πλευρά του ωκεανού. Επίσης η διαθυσιμότητα και η ακρίβεια του να υπάρχουν πολύ περισσότεροι δορυφόροι μπορεί να βοηθήσει την απόδοση, να την ενισχύσει σε περίπτωση που κάποιο σύστημα υπολειτουργεί. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να τονίσω είναι ότι ο Γαλιλαίο, όπως και το GPS, δίνει συγκεκριμένα σήματα τα οποία λαμβάνονται και θεωρούνται ισχυρά σε ό,τι αφορά το μπλοκάρισμα. Είναι δηλαδή σχεδιασμένο ειδικά για να ανθίσταται σε κακές, ε, βλαβερές, επιζήμιες επιθέσεις. Μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε έτσι την ανθεκτικότητα του συστήματος. Και τέλος, και εξίσου σημαντικό, ο Γκαλιλαίο και το έγνος, και ειδικά το έγνος, έχουν σχεδιαστεί για ε, υπηρεσίες ε, κρίσιμες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς, να δίνουν αξιοπρεπείς αξιόπιστες πληροφορίες. Αν μια υπηρεσία δεν είναι αξιόπιστη, αν υπάρχει δηλαδή μια, κακή λειτουργία, τότε μέσα σε 6 δευτερόλεπτα μπορεί ο χρήστη να πληροφορηθεί ότι δεν, το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε μπορεί να αλλάξει και να χρησιμοποιήσει άλλο σύστημα. Να πω λοιπόν απλώς ότι το να εξαρτάται κανείς από ένα σύστημα προφανώς σημαίνει ότι είναι, δεν υπάρχει πολύ περιθώριο α, ε, ε, μανούβρας και χειρισμών, αλλά η δυνατότητα του GNSS προβλέπει αυτή ακριβώς την εξασφάλιση. Το σύστημα θα είναι λειτουργικό. Ε, ευχαριστούμε κύριος Κλάους Χέρμπερτ Ρόλφ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είναι πολύ το σωστό αυτό που λέτε. Στη δική σας τη χώρα αρχές του 2000 ε, εγώ πήγα και μάλιστα υπήρχαν ε, πάρα πολλοί νέοι τότε που προφανώς τώρα θα έχουν μεγαλώσει και ασχολούνται με το θέμα αυτό. Όντως στην χώρα σας έχετε προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν είπα όμως ότι θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τον Γαλιλαίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήδη από τώρα όλα τα μεγάλα συστήματα δορυφόρων. Αυτό που θέλω να πω όμως και ίσως είναι πιο σημαντικό είναι ότι το θέμα που θέτετε, το ερώτημα που θέσατε είναι πού ακριβώς είναι η διαφορά. Για μας ως εταιρεία δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει, το μόνο ζήτημα είναι το θέμα του κόστους. Αλλά αν θέλουμε μια ευρωπαϊκή τεχνολογία ε, δορυφόρων, πρέπει, εφόσον έχουμε τεχνολογία, να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό το κάνουμε με το έγνος ήδη. Περιμέναμε τον Καλιλαίο, περιμένουμε τον Κοπέρνικο να είναι λειτουργικά. Οπότε το ερώτημά σας σωστό είναι γιατί είναι καλύτερο. Χρησιμοποιούμε τεχνική, δεν είναι καλύτερο, ε, χρησιμοποιούμε τεχνική που ήδη υπάρχει. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να έρθουμε στις δικές σας τι μεγάλες ε, εκτάσεις και καλλιέργειες με ένα πρωτότυπο. Χρειαζόμαστε σταθερά συστήματα. Και τι έχει κάνει ο Γαλιλαίο μέχρι τώρα. Στα πρώτα χρόνια, γιατί εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, στα πρώτα χρόνια είχαμε το GPS. Το ε, GPS ε, μπορούσε να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Μπορεί να είχαμε ας πούμε, μια απόκληση ένα, δύο, τέσσερα μέτρα. Από τότε που έγινε όμως το Γαλιλαίο έγινε και το GPS πιο σταθερό. Ε, κατά τύχη έγινε επίτηδες, έγινε δεν ξέρω, αλλά δώστε μας την δυνατότητα να λειτουργήσουμε με ένα ευρωπαϊκό σύστημα, γιατί όντως θα μας είναι χρήσιμο. Ευχαριστώ. Κυρία Νίμπλερ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι όντως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να λειτουργήσει ο Γαλιλαίο και στο Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια το υποστηρίζουμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Έχουν υπάρξει πολλές ε, συζητήσεις και για τη χρηματοδότηση του συστήματος, αλλά το θέμα είναι να παραμείνει η εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε δυνατές ε, ε, υπηρεσίες, να μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας ισχυρές υπηρεσίες για να μπορέσουν να ωφεληθούν. Και ένα δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ιστορικών ασχολούνται με το σκάνδαλο της NSA και την ανεξαρτησία από άλλες μεγάλες ε, παγκόσμιες δυνάμεις μέσω ενός συστήματος ε, δορυφόρων. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και μας απασχολεί και εμάς ως βουλευτές λοιπόν. Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Θα, βάλουμε όλοι μας τη δύναμη, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να εφαρμοστεί, να έρθει στην ε, αγορά. Μιλούμε πάντα για τη χρηματοδότηση. Το, Γαλιλαίο, το θέμα ήταν αν ο Γαλιλαίο θα προχωρήσει ή όχι. Η Κομισιόν έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Τα κράτη-μέλη ήθελαν να μπορούν να ρυθμίσουν τη χρηματοδότηση ε, εθνικά, αλλά εμεί είπαμε ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και έτσι η εμπειρογνωμοσύνη και το αποτέλεσμα δεν θα είναι μόνο για ένα κράτο μέλο, θα είναι κοινό για όλα τα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Ένα τελευταίο ερώτημα ε, για το δεύτερο πάνελ. Ο κύριος Ζητορίδης είπε ότι το η GSA είναι ο εταίρος σας ε, που θα, εξε, που θα εκμεταλλευτεί, που θα αξιοποιήσει τον Γαλιλαίο. Το θέμα των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι ένα θέμα που εσείς ως υπηρεσία παρακολουθείτε. Υπάρχουν μήπως προβλήματα ως προς αυτό, την πνευματική ιδιοκτησία... Ε, γιατί είναι και θέμα που θα απασχολήσει και το δεύτερο πάνελ μας. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτό το θέμα με όσους ε, συνεργάζεστε. Τελευταίες απαντήσεις γιατί μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Μάλιστα. Η ερώτηση για το IPR και πιο συγκεκριμένα για την πολιτική του IPR είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε σήμερα. Ωστόσο δεν είναι άμεσα άμεση ευθύνη της υπηρεσίας. Πρόκειται για μια πολιτική που είναι υπό ανάπτυξη. Όμως επειδή η υπηρεσία μας είναι κοντά στην αγορά συμβάλλει σημαντικά. Φυσικά το συμφέρον μας ε, είναι να προστατεύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει φυσικά να το, να το φροντίσουμε τώρα που ξεκινάμε την εμπορική φάση και έτσι σίγουρα ε, συμμετέχουμε στον καθορισμό της πολιτικής αυτής από κοινού με την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πραγματικά τους δύο εισηγητές. Ολοκληρώσαμε έτσι αυτό το πρώτο τμήμα της ε, συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ και τώρα ζητώ από την ε, Κατερίνη Καβαδά και τον Τζαν Σάρλ Ουρκάντα να ε, λάβουν θέσεις. Ξεκινήσουμε λοιπόν το δεύτερο πάνελ της δημόσιας ακροασής μας, πνευματικά δικαιώματα, δυνατότητες και μελλοντικές εξελίξεις. Το λόγο έχει η κυρία Εκατερίνη Καβαντά, η οποία είναι επικεφαλής του τμήματος ε, δημοσιονομικών θεσμικών ε, θεμάτων και νομικών θεμάτων όσον αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Σας ευχαριστώ κύριε Σαρτόρη. Καλημέρα σε όλους. Καλημερίζω και τους διερμηνείς. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και την ικανοποίησή μας για τη διοργάνωση της σημερινής μικρής δημόσιας ακρόασης. Όπως είπε η κυρία Νίμπλερ, έχουμε την εντύπωση ότι καθότι το 2014 έρχεται μέσα σε λίγους μόνους μήνες, θα πρέπει να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, προκειμένου να καταφέρουμε να αποφεληθούμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βέβαια και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που θα έχουμε. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα σημαντικό το στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματός μας. Εμείς επενδύουμε στο πρόγραμμα αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια και τα IPR αποτελούν πραγματικά απόδοση της επένδυσης αυτής, μια σημαντικότατη απόδοση. Θεωρούμε ότι ως προγραμματιστές, ότι ως διαχειριστές των προγραμμάτων αυτών, αν καταφέρουμε να διαχειριστούμε και να πλαισώσουμε σωστά τα IPR και να τα χειριστούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τότε θα έχουμε μια πολύ μεγάλη χρήση των συστήματών μας σε παγκόσμια βάση και θα έχουμε δεύτερον τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες μας, όχι μόνο την τεχνολογία Γκαλιλαίο, αλλά και τις επιμέρους τεχνολογίες που θα προκύψουν, κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις βιομηχανίες ευρωπαϊκές και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα καταφέρουμε επίσης να συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Υπήρου μας. Όπως είπε ο κύριος Χόρκ, θα μπορούσα να μιλήσω για ολόκληρε ημέρε για το ζήτημα αυτό, αλλά καθότι έχω στη διάθεσή μου μόνο 10 λεπτά, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία κυρίως, σε τρεις κυρίως πτυχές. Η πρώτη έχει να κάνει με το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να αναλάβει δράση όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομικό αυτό πλαίσιο. Δεύτερον θα προσπαθήσω να δω μαζί σας και να σας καταστήσω σαφές ποιες είναι ε, οι βασικοί, οι βασικοί στόχοι πολιτικής και οι βασικές αρχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης κατά την ε, εκπόνηση μιας στρατηγικής πνευματικών δικαιωμάτων. Γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εργαζόμαστε και να μιλάμε για τον Καλλιλέο αν δεν καταφέρουμε να θεσπίσουμε ένα συνεκτικό, σταθερό, ξεκάθαρο πλαίσιο και μια ξεκάθαρη στρατηγική στο ζήτημα αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων. Επ' αυτού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά υποστήριξη και πολιτική καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέλος, θα σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα το οποίο προτίθεται να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη φορά με συγκεκριμένε προτάσεις και ιδέες και όλα αυτά στις αρχές του 2014. Όσον αφορά το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως ξέρετε από το 2008 και μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έλαβαν μια επαναστατική πολιτική απόφαση, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επιτέλους να έχει στην κατοχή της ένα σύστημα, καθώς επίσης και όλα τα υλικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στο σύστημα αυτό. Μέχρι το 2008 Ελάχιστα στοιχεία έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως κάποιους δορυφόρους και βάσεις εκτόκτευσης. Από το 2008 και μετά έχουμε όλη αυτή την ευφυΐα επίσης στην κατοχή μας, δηλαδή πνευματικά δικαιώματα για ό,τι έχει προκύψει από τη δορυφορική έρευνα από το 2008 μέχρι σήμερα. Ήταν επαναστατική απόφαση αυτή για δύο λόγους. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων των σημαντικών στοιχείων του συστήματος Γαλιλαίου. Δεν θα ήταν σοβαρό και επαγγελματικό από τη δική μας την πλευρά να βασιζόμαστε μόνο σε συμφωνίες αδειοδότησης με εμπορικού εταίρους και να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό. Αν κάναμε κάτι τέτοιο θα ήμασταν ποτέ σε θέση να εξασφαλίσουμε την συνέχεια των υπηρεσιών μας. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η υπόφαση είναι επαναστατική είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στην κατοχή της τα κρίσιμα αυτά πνευματικά δικαιώματα, IPR, θα είμαστε σε θέση να έχουμε μία ανοιχτή δωρεάν και ανοιχτή προς όλους πρόσβαση στην τεχνολογία GNSS. Εργαζόμαστε λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους χρήστες εκείνους οι οποίοι θα προσελκυθούν από την τεχνολογία την οποία κατέχουμε και θα επιθυμήσουν να τη χρησιμοποιήσουν. Κυρία Πρόεδρε, προκειμένου να μπορείτε να παρακολουθήσετε καλύτερα την παρουσίασή μου θα έπρεπε να προβάλλουμε και τις διαφάνειες. Παρακαλώ πολύ, βρίσκομαι στην τρίτη διαφάνεια αυτή τη στιγμή. θα παρουσιάσουμε λίγο αργότερα μέσω της παρουσίας του κυρίου Ουρκάντ ποιο είναι το πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων το οποίο έχουμε στα πλαίσια του GNSS. Πρέπει να σας πω ότι ε, τα βασικά πνευματικά δικαιώματα, IP αυτή τη στιγμή, βρίσκονται στην κατοχή της ΚΝΕΣ στη Γαλλία και της ΕΖΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα χαρτοφυλάκιο πνευματικών δικαιωμάτων μικρό αυτή τη στιγμή, το οποίο πρόκειται όμως να αυξηθεί στο μέλλον. Από το 2014 και μετά θα έχουμε μια μεταφορά πνευματικών δικαιωμάτων, κυρίω από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μεταφερθούν δηλαδή όλα τα διπλώματα βρεσιτεχνία προ εμά και θα έχουμε επίση και τη φάση εκμετάλλευση. Και από τη φάση αυτή θα προκύψουν πάλι πνευματικά δικαιώματα τα οποία θα βρίσκονται στην απόλυτη πλέον κατοχή και προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. θα αναφερθώ στο καθεστώς των ανοιχτών υπηρεσιών ICD ένα έγγραφο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο υποστηρίζουν έξι διπλώματα ευρεσιτεχνία, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα. Οι πληροφορίε είναι διαθέσιμε επίση στην ιστοσελίδα μα και πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε κατασκευαστέ παγκοσμίω, σε δωρεάν εντελώ βάση, να έχουν πρόσβαση σε όλε τι τεχνικέ πτυχέ τη διεπαφή ανοιχτή υπηρεσία, Open Service Interface, όπω αυτή προβλέπεται στα πλαίσια του Γκαλιλαίου. από την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα είμαστε σε θέση να έχουμε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι ίδιες αρχές θα ισχύουν και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα δικαιώματα κυριότητας. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε να επεξεργαστεί ένα πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υπάρχουν όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ποιες είναι τώρα οι κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά το πολιτικό αυτό πλαίσιο. Καταρχάς, έχουμε τέσσερις τέτοιες βασικές αρχές. Ο πρώτος στόχος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διασφαλίσει την αρμονική ανάπτυξη της αγοράς GNSS, περιορίζοντας και καταρρύπτοντας όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στην πρόσβαση σε διάφορες κατηγορίες. Όλα θα πρέπει να αναπτύσσονται με τρόπο εναρμονισμένο. Ο δεύτερος πολιτικός στόχος είναι ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο να αναπτυχθούν περισσότερο οι νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει επίσης να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και πρέπει να ενθαρρύνουμε τρίτα μέρη και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι πολύ βασικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτος μας πολιτικός στόχος είναι να προστατεύσουμε και να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στα πνευματικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, αλεξίου σημαντικό, είναι η προστασία των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών. Θα ήθελα να επιμείνω στο σημείο αυτό γιατί όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εργαζόμαστε μεμονωμένα κάθε φορά που μιλάμε για IPR, για πνευματικά δικαιώματα. Δεν είναι δικά μας τα πνευματικά αυτά δικαιώματα, μπορεί εμείς να έχουμε την κατοχή, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρίτοι εταίροι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες, οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και μπορούν να τα αναπτύξουν ακόμα περισσότερο. Τώρα, σε ποια στοιχεία θα βασιστούμε προκειμένου να κάνουμε μία αξιολόγηση της κατάστασης. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία του Γαλιλαίου σε τρίτα μέρη. Εγώ θεωρώ ότι τα όσα κατέχουμε ως γνώση, ως επιρρογνωμοσύνη, θα πρέπει να είναι ανοιχτά προς όλα τα τρίτα μέρη και κατά αναλογία θα πρέπει να έχουμε και κάποιες δυνατότητες αμοιβαιότητας προκειμένου και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε τεχνολογικές εξελίξεις, σε διπλώματα τεχνολογικά ευρεσιτεχνίας τα οποία έχουν αναπτύξει τρίτες εταιρείες, οι εταίροι μας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι όλη αυτή η εργασία την οποία κάνουμε προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες ανεπάρκειες που εντοπίζουμε στην αγορά και να καταφέρουμε να ενθαρρύνουμε μικρομεσαίες και άλλες εταιρείες προκειμένου να καταφέρουν να αναπτύξουν όλα τεχνολογικά αυτά στοιχεία τα οποία θα καταπολεμήσουν τις υφιστάμενες ανεπάρκειες. Επίσης θα πρέπει αυτή τη στιγμή να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο με άλλες πρωτοβουλίες αξιοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να προστατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε περισσότερο τα πνευματικά δικαιώματα. Θα σας παραθέσω τώρα τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε εγκρίνει. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ξεκινήσει μια προπαρασκευαστική εργασία για να εγκρίνουμε το νομοθετικό αυτό ρυθμιστικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να δούμε πόσα διπλώματα βρεσιτεχνίας υπάρχουν στην Ευρώπη, τι ανήκει σε ποιον και ποια διπλώματα βρεσιτεχνίας βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Χρειαζόμαστε μια σφαιρική απογραφή της κατάστασης για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Σε μια δεύτερη φάση θα πρέπει να αναλύσουμε όλες τις πτυχές του φακέλου αυτού σε συνεργασία με όλους τους εμπειρογνώμονες εκπροσώπους της βιομηχανίας και άλλους ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με το παρόν χρονοδιάγραμμά μας, ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι στο πρώτο εξάμεινο του 2014 και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε κατά αυτόν τον τρόπο στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να υποβάλουμε συγκεκριμένες συστάσεις, συγκεκριμένες ιδέες και να παρουσιάσουμε επίσης και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία θα είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά μας και να προωθήσουν περισσότερο τη χρησιμοποίηση του συστήματός μας σε παγκόσμια κλίμακα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κατερίνα Καβαδά. Τώρα το λόγο έχει ο, Ούρκαντ, France Brevet. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτόρη και την κυρία Νίμπλερ από το Ευρωκοινοβούλιο που μου έδωσαν την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις όσον αφορά την διάσταση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των, της ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας που είναι το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Καταρχήν, δύο λόγια Όσον αφορά την France Brevet, πρόκειται για ένα κυρίαρχο, το πρώτο μάλλον κυρίαρχο ταμείο ε, επενδύσεων το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα των ευρεσιτεχνιών. Υπάρχουν τα παρόμοια ταμεία στην ε, Ασία, στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν, στην Κίνα που όλοι έχουν ως ε, σκοπό να βοηθήσουν τα καινοτόμα οικοστήματα στις χώρες αυτές και πιστεύω πως είναι μια ανάγκη που είναι σαφής πλέον δεδομένες της του περίπλοκου χαρακτήρα και της διαχείρισης ε, του θέματος των ευρεσιτεχνιών. Ο στόχος μας, η αποστολή μας είναι πολύ σαφής, να βοηθήσουμε τα δικά μας καινοτόμα οικοσυστήματα, ε, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως, αλλά και τις ε, μικρές, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα, να αξιοποιήσουν από τη μια πλευρά περισσότερο τα αποτελέσματα των ερευνών τους, δηλαδή τα διπλώματα ευρυστεχνίας και να, υπάρχει επιστροφή από τις επενδύσεις, απόδοση των επενδύσεων μέσω ας πούμε των ευρεσιτεχνίων και έπειτα για τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν την ελευθερία ε, εκμετάλλευσης, δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα τα ευρεσιτεχνίας τρίτων και κυρίως τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που δεν είναι ευρωπαϊκά. Αυτά τα δύο προβλήματα συνδέονται απόλυτα, δηλαδή αξιοποίηση και των, των δικαιωμάτων. Στον τομέα της GNSS και του Γαλιλαίου αρχίσαμε να εργαζόμαστε με Ευρωπαίους εταίρους, να συνεργαζόμαστε εδώ και δύο χρόνια περίπου και συνεργαζόμαστε σε, στενά με την ΕΚΝΕΣ στη Γαλλία, με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία αλλά και τους μεγάλους φορείς του τομέα που είναι η EDS, Θαλή, Σαλίνια Space και TomTom. -Tom. Σήμερα θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω μία πρώτη εικόνα για τις αναλύσεις που κάναμε όσον αφορά την κατάσταση πρόοδου. Ποια είναι δηλαδή, ποιο είναι το τοπίο στον τομέα GNSS και Γαλιλαίο, να εντοπίσουμε τους κινδύνους και έπειτα ε, και τις ε, δυνατότητες και κάποιες οδούς για πρόοδο που θα θέλαμε να προτείνουμε. Καταρχήν όσον αφορά το τοπίο, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε το σύνολο των ε, υπαρχών των ευρεσιτεχνιών που δυνητικά είναι εφαρμοστές για το Γαλιλαίο. Στο επίπεδο ε, των υποδομών και των εξοπλισμών έχουμε αναλύσει 2.500 οικογένειες ευρεσιτεχνιών αρκετά σημαντικός αριθμός και έχουμε διαπιστώσει ότι ανάμεσα στις 2.500 αυτές οι οικογένειες οι 26 είναι απολύτως απαραίτητες. Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του Γαλιλαίου. Είναι πιθανόν να υπάρχουν και περισσότερες. Αλλά Αυτό που ξέρουμε είναι ότι 26 από αυτές είναι απαραίτητες. Τώρα, όσον αφορά τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες, εδώ έχουμε εντοπίσει 400 οικογένειες ευρεσιτεχνιών που είτε είναι πολύ σημαντικές είτε απαραίτητες για ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών. Το καλό νέο εδώ είναι ότι το 60% αυτών των σημαντικών ευρεσιτεχνιών είναι στα χέρια ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών ε, ε, ε, εταιριών. Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό και το πολύ θετικό. Ε, τονίζει στον τομέα της ε, πλοήγησης μέσω δορυφόρου τις επενδύσεις που έγιναν από την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες ή δεκαπενταετία μάλλον ε, εξαιρετικού τύπου επενδύσεις και που ευτυχώς μεταφράζονται αυτή τη στιγμή από την ύπαρξη μάλλον την ιδιοκτησία ενός πολύ μεγάλου τμήματος ευρεσιτεχνιών. Ένα στοιχείο πάρα πολύ θετικό. Σημαίνει την αποκριστάλωση αυτής της προσπάθειας επενδύσεων που κατέβαλαν τα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία. 35% ε, των ευρεσιτεχνιών ανήκουν στα αμερικανικές εταιρείες και το υπόλοιπο, ε, αλλά πολύ μικρότερο βέβαια ποσοστό, είναι αυτό που κατέχουν οι ε, κινέζικες εταιρείες. Τώρα, 65% αυτών των ευρεσιτεχνιών ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής δεν έχουν υποχρεωτικά δεσμευθεί όσον αφορά τη διάθεση αυτών των ευρεσιτεχνιών. Από, δεν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι όροι για την χρήση, ε, μάλλον για την θέση στη διάθεσή μας ε, αυτών των ευρεσιτεχνιών, κυρίως από τις μη ευρωπαϊκές εταιρείες, δεν είναι κάτι το δεδομένο. Οι κίνδυνοι λοιπόν είναι αρκετά σαφείς. Ο πρώτος κίνδυνος είναι, και αυτό το ξέρουμε και από πείρα, πως δεν είναι βέβαιο ότι το σύνολο των απαραίτητων ευρεσιτεχνιών για την εφαρμογή του Γαλιλαίου, τόσο όσον αφορά την τον εξοπλισμό αλλά και τις υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμος σε, ο, σε ε, υπό όρους το Στο παρελθόν είδαμε για άλλες τεχνολογίες ε, να μπλοκάρονται λόγω ακριβώς ε, το ότι κάποιες επιχειρήσεις για υπεράσπιση των δικών τους συμφερόντων δεν επιθυμούσαν να τις διαθέσουν ή έθεταν όρους που δεν μπορούσαμε εμείς να ανταποκριθούμε. Έπειτα, 50% των ευρεσιτεχνιών που εξετάζουμε στην ουσία ισχύουν και εφαρμόζονται όχι μόνο για το Γαλιλαίο αλλά και για τα άλλα συστήματα GNSS όπως το GPS 3. 50% δηλαδή των ευρεσιτεχνιών καλύπτουν τόσο το σύστημα Γαλιλαίο όσο και το GPS 3 και σε μεγάλο βαθμό και το μη αμερικανικό ή μη ευρωπαϊκό σύστημα όπως το, το GLONASS που είναι το ρωσικό και το Baidu που είναι το κινέζικο. Εντάξει, είναι και εντυπωσιακό αυτό, γιατί οι βασικές τεχνολογίες είναι συχνά οι ίδιες τα μεγάλα αυτά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί. Αυτό το σημείο ότι δηλαδή αυτά οι σύμβερες τεχνίες χρησιμοποιούνται, είναι κοινέ για όλα τα συστήματα GNSS μπορεί να είναι θετικό αλλά μπορεί να είναι και αρνητικό στοιχείο. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να μπλοκαριστούν κάποιες από τις λειτουργικές από τις λειτουργίες του συστήματος GNSS. Τώρα, με βάση όλα αυτά, Θεωρούμε πως υπάρχουν κάποιες ε, οδοί για προβληματισμό και κάποιες συστάσεις που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Η πρώτη είναι σε απόλυτα, απόλυτη συμφωνία και στηρίζεται και από τον ε, Καναδά ότι στηρίζουμε απόλυτα τον ορισμό μιας στρατηγικής περί πνευματικών ιδιοκτησία, ιδιοκτησίας, μιας γενικής στρατηγικής που από τη μια πλευρά θα έχει στόχο να ευνοήσει και να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή υιοθέτηση και χρήση του Γαλιλαίου. και άρα την επιτυχία του, αλλά και επίσης, και αυτό φυσικά είναι απόλυτα συμβατό, την πρόθεση των φορέων του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος που έχει επιτρέψει και θα συνεχίσει να επιτρέπει την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Προστασία και προώθηση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος. Δεύτερη σημαντική σύσταση στην οποία ε, Εμεί έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους μας ε, τους βιομηχανικούς εταίρους. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία στηρίζεται και θέλει να εξασφαλίσει την ελευθερία χρήσης, δηλαδή την πρόσβαση των Ευρωπαίων φορέων στο σύνολο των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας τα οποία χρειάζονται και ταυτόχρονα την εξασφάλιση και τη βελτιστοποίηση δεδομένης της ισχυρής βάσης ε, των ε, ευρεσιτεχνών που υπάρχουν, υπάρχει μια απόδοση όσον αφορά αυτού του φορείς έρευνα, στις διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να γίνουν, όπως έχει γίνει και σε πάρα πολλού άλλου βιομηχανικού τομείς, διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να γίνουν ανάμεσα στους κατόχους των ευρεσιτεχνιών, των Ευρωπαίων, των Αμερικανών και των Κινέζων. Αυτές ε, οι πρωτοβουλίες ε, θα είναι καλό να συντονιστούν με φύ τρόπο ώστε η ε, βιομηχανία να μπορεί να στηριχτεί στις γενικότερες συστάσεις που θα καθοριστούν και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος συνάδελφος θέλει το λόγο, η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, και οι δύο παρουσιάσεις. Μας δείξατε όντως ότι από το 2014 θα περιμένουμε μια ανακοίνωση για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οπότε νομίζω ότι και εμείς θα την δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το θέμα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων και των ε, ε, των πατεντών ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. όντω. Ε, έχω ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που υπάρχει στον ορίζοντα 2020, αυτό που έχει αποφασιστεί είναι τελεσίδικο είναι το μέτρο, είναι το, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και μπρο ε, τα διπλώματα ευρεστιχνίας ή πρέπει να ξανασκεφτούμε κάτι. Χρειαζόμαστε φυσικά κάποια δικαιώματα για να είναι λειτουργικό το σύστημα, για να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις ε, υπηρεσίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς ο θεσμός που θα έχει χρηματοδοτήσει αυτό το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχει και τον έλεγχό του. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό συγκεκριμένα. Οι κανόνες στον ορίζοντα 2020 είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε από εδώ και ή υπάρχει και άλλος τρόπος να το σκεφτούμε. Ευχαριστούμε κύριος Κάντσιαν. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους πόρους, τους ελάχιστους πόρους που διαθέτουμε. Από τη μία πλευρά βλέπω ότι από την ε, νομοθεσία πλέον τα νέα μέτρα έχουμε ένα πραγματικό άλμα ποιότητος ε, και ευτυχώς βλέπουμε ότι ε, όλα πλέον τυχαίνουν πάρα πολύ καλού ελέγχου. Επομένως, ε, ελέγχουμε ακριβώς ποιος έχει πρόσβαση, ότι η πρόσβαση αυτή είναι δωρεάν, ότι όλοι μπορούν να αποφεληθούν της τεχνολογίας και αυτό είναι θετικό. Από την άλλη μιλάμε όμως και για την απόδοση των επενδύσεων. Ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε και κάποιο κίνητρο όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου και αυτός να προσελκυθεί και να συμβάλλει στους λίγους πόρους που εμείς έχουμε με τους δικούς του πόρους. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω το εξής. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Όσον αφορά όμως τις μελλοντικέ εξελίξεις, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν με λίγα χρήματα. Μπορούμε πραγματικά να εφαρμόσουμε μια πολιτική εταιρική σχέση ιδιωτικού δημοσίου τομέα στις συνθήκες αυτές προκειμένου να καταφέρουμε το συντομότερο δυνατό να καταλήξουμε στη δημιουργία των εφαρμογών αυτών οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν το συντομότερο δυνατό ή ενδεχομένως να επηρεαστούμε αρνητικά από τους λίγους πόρους που έχουμε. Ουσιαστικά πιστεύετε πραγματικά ότι έχουμε δυνατότητες για να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί σίγουρα ορισμένα πράγματα έχουν επιτευχθεί, αλλά νομίζω ότι καταβάλλονται πάρα πολλές προσπάθειες αυτή τη στιγμή και πολλές φορές δεν καταφέρνουμε τελικά στην πράξη να ενεργοποιήσουμε τη συμπράξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Πρόεδρος, υπάρχει κανείς άλλος που θέλει το λόγο, δεν νομίζω. Επομένως, σας ακούσουμε για μία πρώτη απάντηση την κυρία Καβαδά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. να απαντήσω πρώτα στην ερώτηση της κυρίας Νίμπλερ. Ο, τον Γαλιλαίο χρηματοδοτείται καταρχάς από τον προπολογισμό GNSS, όπου υπάρχει εδώ πέρα μια συγκεκριμένη πολιτική χρηματοδότηση στα πλαίσια του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και όσον αφορά τις συγκεκριμένες εφαρμογές, λαμβάνουμε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Και όπως πολύ σωστά είπατε, υφίσταται ήδη ένα πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει και προωθεί την πολιτική IPR για τα πνευματικά δικαιώματα. Εμείς με το δικό μας νομοθετικό κείμενο θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε δύο συγκεκριμένες βάσεις οι οποίες να μην αντιτίθενται η μία στην άλλη και να μην τίθενται καντά των βασικών αρχών και των βασικών στοιχείων του προγράμματος. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε με το νέο κείμενο, το οποίο όπως είπα θα φτάσει το 2014 στο Κοινοβούλιο, είναι να επιτελέσουμε ένα βήμα πρόοδου. Να λέμε ότι δεν θα υπάρχει διαφορετικό σύστημα κυριότητας για κάθε ξεχωριστό πρόγραμμα στα πλαίσια του GNSS, θέλουμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εναρμονίσουμε τους δύο αυτούς τομείς και πώς θα καταφέρουμε να εμπλέξουμε και άλλους παράγοντες και άλλους φορείς όσον αφορά στην κυριότητα αυτών των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Τώρα όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση και τη νομική πτυχή. Σίγουρα η πνευματική κυριότητα είναι κάτι το οποίο κοστίζει. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να δούμε πώς θα καταφέρουμε με έναν ισορροπημένο τρόπο να επιμερίσουμε όλο αυτό το κόστος και πώς θα μπορέσει το κόστος αυτό να, να μεταφραστεί σε όφελος και κέρδος για την Ευρώπη. Δεν θέλουμε απλώς εμείς να επεξεργαστούμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα δικά μας. Θέλουμε θέλουμε να καταφέρουμε να αποφεληθούμε και από τα υπόλοιπα διπλώματα ευρεσιτεχνία τα οποία έχουν αναπτυχθεί από άλλε εταιρείε και άλλου φορεί στην Ευρώπη. Είδαμε και από την παρουσίαση του κυρίου Ουρκάντ ότι υπάρχει μια κοινή βάση εργασίας αυτή τη στιγμή και όπως άλλοι υποφελούνται από εμά, έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποφεληθούμε από τις ευρεσιτεχνίες άλλων. Τώρα, όσον αφορά τα PPP, τις εταιρικές σχέσεις δημοσίου-δημόσιο τομέα, να πω το ακόλουθο. Πριν από μερικά χρόνια, όταν επεξεργαζόμασταν περισσότερο την ιδέα αυτή του PPP, συντοπίσαμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους της αποτυχίας του ήταν ο κίνδυνος στην αγορά. Δηλαδή, εκείνη την εποχή, κανείς και τουλάχιστον οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που είχαν κληθεί να επενδύσουν, δεν είχαν δει αν πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες αγοράς, αγορές εκμετάλλευσης δηλαδή των τεχνολογιών αυτών. Αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δημιουργήσει νέες τεχνικές εφαρμογές, ένα νέο σταθερό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου μπορούμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα, μπορεί αυτό να εγκριθεί από τους χρήστες και κατά αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος στο πλαίσιο της αγοράς μειώνεται ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε μερικά χρόνια ο κίνδυνος αυτός θα είναι πλέον ελκυστικός αν θέλετε για διάφορες επιχειρήσεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν και σε συνεργασία με το σύστημα για τα πνευματικά δικαιώματα να προσελκύσουμε περισσότερους φορείς από την ιδιωτικό τομέα. Προς αυτό το στόχο ουσιαστικά εργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο Ζαν Κάντε θέλει να πάρει το λόγο. Νομίζω ότι ε, η επόμενη φάση θα είναι σημαντική και χαίρομαι όλους ιδιαιτέρως που βλέπω ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται και προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλαίσιο προκειμένου να καταφέρουμε από τώρα μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2014 να έχουμε μια σφαιρική πλέον εικόνα και να καταφέρουμε να διορθώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και τις πρωτοβουλίες του βιομηχανικού τομέα. Νομίζω ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας αρκεί και θα μας επιτρέψει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες συζητήσεις, να ακούσουμε όλους εμπλεκόμενους εταίρους και φορείς, να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες οι οποίες όντως υφίστανται και είναι πολύ σημαντικές, ευκαιρίες δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση όλων αυτών των σημαντικότατων επενδύσεων που έχουν γίνει, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και το οποίο στην πράξη θα πάρει τη μορφή της βάσης αυτής πολύ σημαντικών ευρεσιτεχνιών. Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε και τις ευκαιρίες αλλά και τον κίνδυνο Ξέρετε ότι ζούμε σε έναν πολύπλευρο κόσμο, επομένως θα πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι σχέσεις μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά μια τεχνολογία η οποία εκφύσεως είναι παγκόσμια. Και πέρα από όλα αυτά θα πρέπει επίσης να πετύχουμε την κατάλληλη δυνατή ισορροπία έτσι ώστε και να διασφαλίσουμε την επιτυχία του προγράμματος και την πλήρη εφαρμογή της τεχνολογίας Γκαλιλαίου Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για το ζήτημα αυτό και από την άλλη βέβαια να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση επενδύσεων και ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή ανταγωνιστική θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς φορείς σε έναν ανταγωνισμό, σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού που είναι πλέον παγκόσμιο. Και ευχαριστούμε η Αντζέλικα. Θέλει να πει κάτι ακόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο φράσεις μόνο. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους ομιλητές μας στο δεύτερο πάνελ και δύο φράσεις έτσι συνοψίζοντας ε, από όσα μπορώ να συμπεράνω από την ε, ακρόασή μας σήμερα το πρωί. Νομίζω καταρχάς ότι το αποτέλεσμα του πρώτου πάνελ ήταν ότι πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η τεχνογνωσία θα πρέπει να παραμείνει εντός Ευρώπης. Ε, το λέω έτσι πολύ συγκεκριμένα, από ένα ευρώ πρέπει να μπορούμε να βγάλουμε δέκα ευρώ. Ε, αν τα πράγματα λοιπόν πάνε καλά θα μπορέσουμε να δεκαπλασιάσουμε τις επενδύσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό μήνυμα να βγει. Επίσης ε, το έγνος και τον Καλιλαίο είναι αρκετά, ε, θα είναι αρκετά λειτουργικά. Ε, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη για αυτά τα συστήματα. Έχουμε και τις εκλογές βέβαια την επόμενη χρονιά, οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα ότι θα υπάρξει κάτι που θα βοηθήσει τους ανθρώπους, έστω και αν αυτό το κάτι βρίσκεται στο διάστημα. Χάρηκα που άκουσα από τον κύριο Ρόλφ τα όσα μας είπε για την έξυπνη γεωργία, πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Καλλιλέο και τον Κοπέρνικου για την γεωργία, για τι καλλιέργειε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη-μέλη μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Επίση, Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακούσαμε και για του κινδύνου που μπορεί να υπάρξουν. Η σταθερότητα του συστήματο είναι κάτι που πρέπει να μπορούμε να το εγγυηθούμε και στο GSA θα πρέπει να κάνουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να μείνουν τα πράγματα σταθερά και βεβαίως έχουμε το θέμα και της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημά μας να είναι αξιόπιστο όπως είναι το GPS και όπως είναι και τα υπόλοιπα. Ακούσαμε λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από το πρώτο και από το δεύτερο πάνελ. οι αριθμοί που μας αναφέρατε εσείς ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για τον Καλλιλέο, για τον GNSS, για τις υπηρεσίες που θα μπορέσουν να προκύψουν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βεβαίως χαίρομαι που διαπιστώνω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή σε ό,τι αφορά τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Νομίζω το μήνυμα που βγαίνει από αυτό είναι ότι μπορεί να υπάρχουν μεν κίνδυνοι, αλλά έγκαιρα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική, κυρία Καβαδά, η οποία θα εξασφαλίζει τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Νομίζω ότι και αυτό σε πολιτικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό. Είπατε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει απόλυτο έλεγχο του συστήματος, δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εκεί τίθεται και το ερώτημα των δικαιωμάτων ε, που είναι κάτι ουσιώδου σημασίας. Επίσης ελεύθερη πρόσβαση, ε, απάλληψη της διακριτικής μεταχείρισης. Ε, θα περιμένουμε από εσάς την ανακοίνωση ε, το 2014 για να δούμε πώς μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, του κινδύνους, πώς μπορούμε να τους ελαχιστοποιήσουμε. Σας λέω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ όλους που ήρθατε και είχαμε μια, πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ε, να συνεχίσουμε και τον επόμενο χρόνο ε, τέτοιες ενδιαφέρουσες ακροάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ, την Κατερίνη Καβαδέ και τον Ζαν Σάρλο Ουρκάντε, ολοκληρώσαμε έτσι και αυτό το δεύτερο πάνελ. Για τα συμπεράσματα, τώρα στις 10.30 και 35 μάλλον, θα πρέπει να έρθει ο Επίτροπος Ταγιάννη, ο οποίος ελπίζω θα μας δώσει, α, μάλλον να πω, ελπίζω σωστές πληροφορίες θα έχει φύγει εδώ και λίγα λεπτά και έρχεται από την Κομισιόν. Αν αποφασίσουμε λοιπόν να περιμένουμε τον Επίτροπο, έχουμε 10 λεπτά, 8 λεπτά διάλειμμα για έναν καφεδάκι μέχρι να φτάσει ο Επίτροπος. και δεν Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ παρόντες. Να ευχαριστήσω επίσης τους προσκεκλημένους μας που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Ταγιάννη, ο οποίος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθότι συνεδρίαζε το Σώμα των Επιτρόπων. Όπως γνωρίζει ο Επίτροπος, έλαβε χώρα μια συζήτηση με δύο πάνελ για ζητήματα τα οποία άπτονται του Γκαλιλαίου. Θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όχι μόνο για την πρόσκλησή σας, αλλά γιατί η Επιτροπή σας αποφάσισε να τονίσει τη σημασία που έχει για την βιομηχανική πολιτική η ε, διαστημική δραστηριότητα και η διαστημική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας ε, το καταπληκτικό αποτέλεσμα που είχαμε στις 24 Ιουλίου όταν ε, είχαμε το πρώτο δημόσιο τεστ, την πρώτη δημόσια δοκιμή λειτουργίας δορυφόρου του Γκαλιλαίου, το οποίο έδωσε πολύ θετικά αποτελέσματα. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη θέση τοποθέτησης του δορυφόρου και να τεθεί αυτός σε συγκεκριμένη τροχιά στο διάστημα. Το αποτέλεσμα αυτό, το επίτευγμα αυτό δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό επιστημονικό επίτευγμα. Είναι και ένα πραγματικό πολιτικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κατέδειξε ότι είναι σε θέση να πετύχει θετικά αποτελέσματα μέσω του GNSS. Μάλιστα τον Καλιλαίο ξεπέρασε ως προς τις α, λειτουργίες του το αμερικανικό GPS και μάλιστα έχει ένα περιθώριο σφάλματος μικρότερο από τα δύο μέτρα. Αυτό ξεπέρασε κάθε αναμονή βασικά, γιατί ε, ουσιαστικά βαρσιζόμαστε μόνο στους τέσσερις ε, δορυφόρους οι οποίοι έχουν τεθεί αυτή τη στιγμή σε τροχιά. Κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να έχουμε πολλές νέες υπηρεσίες πέρα από τη δορυφορική πλοήγηση και πέρα από το το κόμπας και όλα τα άλλα δορυφορικά συστήματα τα οποία εφίστανται σήμερα. Και καταλαβαίνετε ότι από αυτό θα αποφεληθούν και οι υπόλοιπε ευρωπαϊκές βιομηχανίες σε άλλους κλάδους δηλαδή. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και θα τα δούμε αυτά και στο διάστημα αλλά και στην επίγεια βιομηχανία. Και όπως είδατε και από τις παρουσιάσεις που ακούσατε, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι θα επωφεληθούν ε, από το σήμα αυτό του Γκαλιλαίου καθώς επίσης και από τη διασταύρωση του σήματος Γκαλιλαίου και Κοπέρνικους και θα καταφέρουμε επίσης να έχουμε και πιο προηγμένες μορφές πολιτικής προστασίας σε περίπτωση θεομηνιών. Χάρη στο Κοπέρνικους καταφέρνουμε και έχουμε μια πολύ καλύτερη παρακολούθηση της γης. Μπορούμε και βλέπουμε ακριβώς που έχουν συμβεί καταστροφές, που πρέπει να επέμβουμε για έρευνα και διάσωση που πρέπει να επέμβουμε με διαφορετικά μέσα. Και το σήμα του Γαλιλαίου θα συνοδεύσει τους διασώστες και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουν αυτοί στα χέρια τους περισσότερα μέσα προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν μια πιο σφαιρική ε, έρευνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πρώτες υπηρεσίες του Γαλιλαίου να είναι διαθέσιμες ήδη από τις ε, αρχές ε, του 2015 και προτού ολοκληρωθεί ουσιαστικά όλο το σύστημα υποδομής, όπως και προβληθεί δηλαδή από την αρχή. Πρόκειται για μια πολιτική προτεραιότητα να καταφέρουμε δηλαδή να εφαρμόσουμε τον Γαλιλαίο πριν ολοκληρωθεί η θητεία, η θητεία μου, η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν γέννη και δηλαδή νωρίτερα από ό,τι απαιτείται για να τεθείουν σε εφαρμογή και σε τροχιά όλοι οι δορυφόροι, όλος αυτός ο αστερισμός των δορυφόρων. Πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ε, επενδυθεί και τον Καλλιλέο θα μας βοηθήσει να καταφέρουμε να έχουμε πρόσβαση σε νέους τομείς της αγοράς και κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφεληθούν πολλές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα καταφέρουμε επίσης να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και θα έχουμε μία επίπτωση της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια ε, βάσει των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχουν επενδυθεί για το Γαλιλαίο. Θα δημιουργηθούν επίσης και πολύ δικευμένες θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ε, καταρχάς ε, στο Λονδίνο και αργότερα σε κάποια άλλη συνεδρίαση ήμασταν σε επαφή με τις εταιρείες εκείνες οι οποίες ε, ασχολούνται με την εφαρμογή στην πράξη όλων των υπηρεσιών που απορρέουν από τον Γαλιλαίο. Με την κυβέρνηση του Μένου Βασιλείου διοργανώσαμε μία διάσκεψη πρόσφατα στο Λονδίνο και μία άλλη διάσκεψη έλαβε χώρα στο Φούλτσινο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Ξέρετε επίσης ότι υπάρχει και μία εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρουμε να καταδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πώς θα χρησιμοποιηθούν και σε τι χρησιμεύουν τελικά τα σήματα του Γαλιλαίου. Ξέρετε ότι στη Ρώμη είχαμε μια τεράστια επιτυχία κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Μέσα σε έξι μέρες 50.000 άτομα επισκέφθηκαν την έκθεση αυτή την οποία ε, Οργάνωση γενική μου διεύθυνση, την οποία θα θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά για το έργο της και για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και ξέρετε ότι κάθε μέρα από τις έξι αυτές μέρες είχε και ένα διαφορετικό θέμα και επέτρεπε στους πολίτες να γνωρίσουν ακριβώς πώς λειτουργεί τον Καλλιλέο και ποιες είναι οι σχετικές υπηρεσίες. Ανάλογη εκδήλωση τώρα θα διοργανωθεί και στο Βίλνιους και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν οι επιχειρήσεις αλλά και οι θύνοντες πολιτικοί από τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι βιομηχανικές εφαρμογές του Γαλιλαίου. Αφού πετύχαμε, μάλλον για να πετύχουμε τους βασικούς αυτούς στόχους, θα πρέπει να προτιμάσουμε κατάλληλα και το έδαφος. Χάρη στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον νέο καονισμό GNSS, που πρόκειται να εγκριθεί τον επόμενο μήνα, χάρη στην χρηματοδότηση που θα δοθεί με ορίζοντα το 2020 μπορούμε πραγματικά να επιτελέσουμε και να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Κατά αυτόν τον τρόπο επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία μελέτη όσον αφορά τις προπτικές της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και κάποια τη δυνατότητα νέων ρυθμιστικών μέτρων προκειμένου τον Γαλιλαίο να εφαρμοστεί στην αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής και δεν αποκλείουμε να έχουμε και μία ρυθμιστική πρόταση ως προς αυτό. Δεν ξεκινάμε, σας είπα, από το μηδέν και θα ήθελα να αναφερθώ στην νομοθετική πρόταση η οποία εγκρίθηκε για το έγνος. Προβλέπετε ότι ε, οι δέκτες οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται πάνω στα αυτοκίνητα για να χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση να δέχονται πλέον το σήμα του Γκαλιλαίου. Και αυτό αποτελεί όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους τους κατασκευαστές δεκτών προκειμένου οι δέκτες αυτοί να είναι συμβατοί με το σήμα του Γκαλιλαίου. Αυτό με τη σειρά του όπως καταλαβαίνετε θα μας ανοίξει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης νέων αγορών. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο να στηρίξει την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για το Κοπέρνικους θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέσω του προγράμματος αυτού να έχουμε μια καλύτερη παρακολούθηση της γης, του περιβάλλοντος και να καταφέρουμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες ασφάλειας. Χάρη στο σήμα του Κοπέρνικους μπορούμε να έχουμε καταπληκτικά αποτελέσματα ακόμα και τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Επομένως θα ενισχυθούν πάρα πολύ όλες οι ομάδες έρευνας και διάσωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δική σας την Επιτροπή που πραγματικά ενέκρινε να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα προγράμματα Κοπέρνικους από τον κοινοτικό προπολογισμό. Θα πρέπει όμως να εγκρίνουμε γρήγορα και το σχετικό καονισμό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθα σε επαφή και ήταν παρούσα και η κυρία Σαρτόρη ο κύριος Πρόντι, καθώς επίσης και κάποιες σκιώδεις ηγητές. Είχα λοιπόν κάποιες επαφές μαζί τους προκειμένου να ακολουθήσουμε μια διαδικασία γρήγορη, fast track. Ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια καθόδη προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε πολύ γρήγορα να καταλήξουμε στη συμφωνία. Τέλος, θα ήθελα να καταφέρουμε να στείλουμε τα σήματα α και β το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητώ και από τη δική μου τη Γενική Διεύθυνση να ακολουθήσει μια διαδικασία fast track και να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν τα δύο αυτά συστήματα. Και καθότι μιλάμε για χρονοδιάγραμμα, θα ήθελα να συνεμερώσω και για το εξή. Κάποια προγράμματα αποφορούν το Γκαλιλαίο. Πριν από μία εβδομάδα συναντήθηκα με τον Ζαν Ζάκ για να μιλήσουμε για την υποδομή και την παροχή υπηρεσιών εντοπισμού θέσης. Ο κύριος Νταρντάν μου είπε ότι ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες από το, κατασκευ... το κατασκευαστή, τον γερμανό κατασκευαστή των δορυφόρων, η ΕΖΑ θα είναι σε θέση να παρουσιάσει επικυρωμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Οκτώβριο. Ο κύριος Νταρντάν επίσης μου είπε ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στις πρώτες υπηρεσίες, οι οποίες όπως, είχαν, όπως είχε προβλεφθεί θα είναι διαθέσιμες στα τέλη 2014 και αρχές 2015. στις επόμενες λοιπόν εβδομάδες, αυτή στιγμή θα έχω στα χέρια μου όλες τις πληροφορίες, θα διοργανώσω μία διοργανική συνεδρίαση για τον Καλλιλέο προκειμένου να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το τελευταίο τελικά, το τελικό χρονοδιάγραμμα το οποίο θα μου δώσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Εν τέλει, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Κοπέρνικους και τον Γαλιλαίο παρέχουν καταπληκτικές ευκαιρίες για τους νέους ερευνητές και τους νέους επιχειρηματίες. Πολλές νέες start-up θα μπορέσουν να προκύψουν χάρη στις εφαρμογές Γαλιλαίου και Κοπέρνικους και θα μπορούσε για παράδειγμα να αναφερθώ στο παράδειγμα μιας νέας ερευνήτριας από το Πανεπιστήμιο Λασαπιέντσα της Ρώμης, το οποίο πήγα και εγώ η οποία δημιούργησε μία νέα λογιστική εφαρμογή για την κωδικοποίηση του σήματος του Γκαλιλαίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και οι ίδιοι έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα προγράμματα αυτά. Το Γαλιλαίο και το Κοπέρνικους θα αποτελέσουν πραγματικά ένα εργαστήριο βιομηχανικής καινοτομίας και έρευνας που θα καταφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουν νέες ευκαιρίες στα ταλέντα, στους νέους μας οι οποίοι έχουν πολύ υψηλή ειδίκευση και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν και αυτοί να συμβάλλουν στην πολιτική ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη μέσω της οποίας θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κρίση, την οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου που θα ασχοληθεί με το ζήτημα της βιομηχανικής πολιτικής θα καταφέρει ελπίζω να ασχοληθεί και με το ζήτημα της ε, διαστημικής πολιτικής και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε όπως έχουμε το Fiscal Compact να έχουμε και ένα Industrial Compact, ένα σύμφωνο δηλαδή για τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πετύχουμε πραγματικά την λεγόμενη επαναβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως άλλωστε ζητάνε και οι τρεις βασικές ομοσπονδίες ε, βιομηχάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία, την Γαλλία και την Ιταλία. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους ιδιαίτερο τη δική σας την Επιτροπή Βιομηχανίας για την υποστήριξή σας και για το ότι προωθείται αυτή τη στιγμή μια νέα βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προωθεί την ανταγωνιστικότητα και σέβεται το περιβάλλον. Ευχαριστώ Επίτροπε. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε τις τακτικές εργασίες της Επιτροπής μας. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, ένα λεπτό ο καθένας, μπορούμε να αφιερώσουμε κάποια λεπτά παραπάνω στην επίσκεψη του Επιτρόπου. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι. Όλοι είναι ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν από τον Επίτροπο, τον οποίο και ευχαριστούμε ακόμη μια φορά και που θα τον έχουμε πάλι εδώ όταν θα το ζητήσει η Επιτροπή και όταν θα θεωρεί, το θεωρήσουμε σκόπιμο να τον καλέσουμε. Σας ευχαριστώ. Bene, iniziamo i lavori della Commissione. Eh, c'è la presente il collega Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Έχουμε την έκθεση του ε, συναδέλφου Φρανκ Προύς που είναι εισηγητής για το CARS 2020. Έχουμε 45 λεπτά προβλέψει για, αυτή την, ε, για αυτό το θέμα, οπότε δίνω αμέσως το λόγο στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει το σχέδιο του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αν μου επιτρέπετε, εξ αρχής θα ήθελα να θέσω σε ένα πλαίσιο ε, την εργασία που μας περιμένει ασχολούμεθα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα θέματα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε CARS 2020. Νομίζω πως αυτό είναι πολύ θετικό γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία απεικονίζει ολόκληρη την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και την κατάσταση των πολιτών. Εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτών και γι' αυτό και θα ήθελα, ε, θέλω πραγματικά να οδηγήσω το Κοινοβούλιο προς ένα κείμενο που θα προσθέσει στη συζήτηση δεν θα έχει βέβαια καμία δεσμευτική αξία το κείμενο αυτό, αλλά γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε απλό, συγκεκριμένο και προσιτό για όλους τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Ως βάση για την έκθεσή μου θα σας πω ότι στόχος ήταν κυρίως να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης, η τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα παραγωγής στην Ευρώπη πριν να αντιμεταρρυθμίσουμε, να ορίσουμε προτεραιότητες και πέρα από τις πολιτικές ιδεολογίες. Η βασική ιδέα είναι να θέσουμε τις πολιτικές μας στην υπηρεσία της καινοτομία, στην υπηρεσία των όσων δημιουργούν, γιατί η καινοτομία αποτελεί το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει στην κατοχή της η Ευρώπη έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Αντί λοιπόν να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, να σκεφτούμε τους τρόπους για να μπορέσουμε να αναζωογονηθούμε. Θα σκεφτούμε όλα, κάπως όπως και οι ΙΠΑ έκαναν για τον τομέα το αυτοκινήτου και δεν διέφυγε ε, κανενός ότι ήταν επιτυχία ε, η προσπάθεια αυτή. Αρχή να δει κανείς τα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει να επηρεαζόμαστε από τους ανταγωνιστές μας ε, ε, και να αποκαλούμεθα όσοι ωραία κοιμωμένοι της, αυτοκινητο, ε, αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα πρέπει να μιλήσουμε όλοι με μια φωνή. Και πριν να σας αναφέρω τους δικούς μου προβληματισμούς, θα ήθελα να σας αναφέρω μια ανησυχητική διαπίστωση που θα πρέπει όμως να διορθωθεί. Η, η υπερπαραγωγικότητα και η αναδιάρθρωση που συχνά είναι οδυνηρές είναι τα δύο βασικά φαινόμενα αυτής της ε, κρίσης ταυτόχρονα είναι συντελεστές και συνέπειες της κρίσης. Ε, θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί αυτές, ε, αυτά όλα επηρεάζουν την, ε, τον κλάδο. Ε, αν δεν μπορέσουμε να τα λάβουμε αυτά υπόψη, πώ θα αποκριθούμε αποτελεσματικά στην κρίση. Θα ήταν σαν ένα ε, γιατρό να προβεί σε διάγνωση χωρί να κροαστεί τον ασθενή. Η κρίση δεν έχει αγγίξει με τον ίδιο τρόπο τους κατασκευαστέ, τα τμήματα τη αγορά, τα προϊόντα ή του διάφορου κλάδου. Αλλά βασικά ορισμένες μάρκες ή κατηγορίε αυτοκινήτων έχουν γλιτώσει από την κρίση, αλλά σήμερα σχεδόν καμιά ευρωπαϊκή εταιρεία δεν είναι καλυμμένοι από την κρίση. Δίνονται βέβαια κάποιες οδηγίες για την έξοδο από την κρίση, όμως θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά με προσοχή, γιατί πρόκειται για προβλέψεις και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη η αγορά, αλλά όλες αυτές οι ωραίες υποσχέσεις θα μείνουν κενό γράμμα, εάν δεν ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των καιρών. Βελτίωση των πολιτικών. Πολιτικός εθελοντισμός χρειάζεται για να υπάρξει μια ατζέντα βραχυπρόθεσμα για δράσεις. Με αυτό το νέο κεφάλαιο το οποίο εγώ εισάγω θέλησα να οδηγήσω όλους να θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα. Πού βρισκόμαστε σήμερα, έχουμε φτάσει στο καλύτερο επίπεδο συντονισμού, έχουμε δώσει τα περισσότερα κίνα μέσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο σε θέματα πολιτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινωνική και φορολογική σύγκληση μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Τι θυσίες θα οφείλουμε να κάνουμε για να τα καταφέρουμε, γιατί να μην εμπνευστούμε από μεθόδους που έχουν λειτουργήσει εδώ, όπως στην αεροναυπηγική στο διάστημα Δεύτερον, να ενισχύσουμε τη θέση μας στις αγορές, είτε τις εσωτερικές είτε τις εξωτερικές. Για την εσωτερική αγορά χρειάζεται να προστατευτούν καλύτερα τα πνευματικά δικαιώματα και τα βιομηχανικά δικαιώματα, καθώς και το απόρριτο το επιχειρησιακό, το επιχειρηματικό, αλλά και οι δοκιμές των προϊόντων πριν να τεθούν σε εμπορία αλλά κυρίως για την εξωτερική αγορά θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε θύματα, να επιβάλλουμε την αμοιβαιότητα στις εμπορικές μας σχέσεις, να ενισχύσουμε το πλωστάσιό μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συμφωνιών, σκεφτόμενοι τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα τομέα. Επιβάλλουμε τις δικές μας προδιαγραφές σε διεθνές επίπεδο, ώστε να μην μας υπαγορεύουν ε, την ε, βιομηχανική τεχνογνωσία και συνοδεύσουμε καλύτερα τις μικρομεσαίες μας προς τον ε, διεθνή στίβο. Η Κομισιόν έκανε πολύ καλές προτάσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας στο χρηματιστήριο νέο είδος χρηματοδότησης όπως οι Business Angels. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της οικονομίας και όχι το αντίστροφο, όπως το κάνουν και οι ανταγωνιστές μας. Σας δώσουμε οξυγόνο στις επιχειρήσεις, κυρίως σε περίοδο κρίσης. Τρίτον, ε, τέταρτον, ας είναι οι κανονισμοί μας πιο δραστήριοι πιο και λιγότερο δεσμευτικοί. Εφηή νομοθεσία λέγεται αυτό και η Κομισιόν το έχει αυτό ε, εμπεδώσει, να ε, εξετάσουμε τις επιπτώσεις όλων των νέων κανονισμών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας Επίσης, οι ρυθμίσεις μας να είναι πιο, απλής, πιο, πιο απλές, πιο κατανοητές, γιατί πολύ συχνά δεν υπάρχει συνοχή και τέλος θα ολοκληρώσω με τη βάση της επιτυχίας μας, δηλαδή τους ανθρώπινους πόρους. Δέχομαι φυσικά θετικά την πρόταση της Κομισιόν, ωστόσο διαπιστώνω πως η αγορά εργασίας δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του τομέα. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων ώστε να προβλέψουμε την αυριανή ζήτηση. Φυσικά πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών, αλλά είναι καθήκον μας να επιμείνουμε για αυτά τα κριτήρια από τη και πρέπει μάλιστα να δεχτούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος στο πλαίσιο των διαφόρων κλάδων και των επιχειρήσεων. Θα σας δώσω, δεν σας δίνω καμιά μαγική λύση. Η Ευρώπη, η Ευρώπη και η Ευρώπη είναι η λύση και το πιστεύω ακράδαντα. Η κρίση είναι εξαιρετικά ισχυρή για να ξεκινήσουμε διχασμένοι. Χρειάζεται να δώσουμε μια κοινή απάντηση και κυρίως σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ώστε να δώσουμε ε, ε, μήνυμά μας. Αυτά τα λόγια είχα να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι και φυσικά περιμένω τώρα τις παρεμβάσεις σας και σε, ένα δεύτερο, σε δεύτερη φάση της τροπολογίας σας. Σας ευχαριστώ. Eh, σας, σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κρέχ. Σας ευχαριστώ. Ισχύει κύριε, δεδομένε τη πολύ άσχημη κατάσταση που διαρκώ επιδεινώνεται στον τομέα τη ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία, ε, η Κομισιόν προτείνει το πρόγραμμα αυτό CARS 2020 ε, είναι μια καλή πρωτοβουλία. Το κόδωνας κινδύνου στον τομέα εξ αρχής ήταν ε, ένα μειούμενη ζήτηση. Από τα 17 εκατομμύρια στα 12 εκατομμύρια έχουμε επεφτάσει το χρόνο. Πώς εξηγείται αυτή η μείωση των, ε, της ζήτησης μόνο λόγω κρίσης. Στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή η τάση είναι η αντίστροφη. Υπάρχει αύξηση από τα 13 στα 17 εκατομμύρια. Αντίθετα στην Ευρώπη η κρίση είναι βαθαίνει όλο ένα. Γιατί γιατί η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη από την, που είναι πολύ μεγαλύτερη από την Αμερικανική, ε, είναι τόσο αδύναμη. Είναι σταθερέ αγορές και οι δύο. βρούμε λοιπόν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Κάποιες απαντήσεις, ε, ε, μάλλον κάποιες προτάσεις έγιναν από τον εισηγητή Προύστου, τον οποίο μάλιστα θα ήθελα και να συγχωρώ για την εξαίρετη εργασία του, αλλά το υλικό που προετοίμασε η Κομισιόν, που ονομάζεται CARS 2020, δυστυχώς περιλαμβάνει βασικά λάθη και κάποιες ε, πολύ λανθασμένες απλουστεύσεις ε, γιατί περιορίζεται στους Ευρωπαίους ε, παραγωγούς και ξεχνά μια πιο γενική προσέγγιση. Ο, αυτο, τομέας αυτοκινητοβιομηχανίας δεν λειτουργεί ξέχωρα. χωρίς δηλαδή όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Η διαρκώς η κρίση βαθαίνει στον τομέα του αυτοκινήτου και μας δείχνει πως η κρίση ευρύτερα στην Ευρώπη δεν προχωρά στο τέλος της. Ε, έχουμε και πάλι να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο, αλλά είναι και μεγαλύτερη ανεργία. Το πρόβλημα είναι ευρύ και είναι πολύ ωραία και καλά αυτά που μας είπε ο Επίτροπος Ταγιάννη που τόνισε την, την, την βούληση να αναπτύξει όλο ένα και περισσότερο την βιομηχανική στρατηγική. Αλλά επανερχόμενη στην έκθεση, ο εισηγητής Προύστου δικαίως και σωστά λέει πως υπάρχει ο κίνδυνος θα ε, ε, λέει ότι θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, τι είναι ευρωπαϊκή επιχείρηση. Πρέπει να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ε, αυτοκινητοβιομηχανία ή όλες τις εταιρείες που λειτουργούν στην επικράτειά μας. Κατά τη γνώμη μου, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν κάποια πολύ δυνατά σημεία στρατηγικές ε, κόστους ε, πολύ θετικές θετικές όπως η στρατηγική της διαφοροποίησης και εδώ έχουμε καλά αποτελέσματα ε, και μια άλλη στρατηγική που δεν είναι και τόσο θετική, είναι πιο δαπανηρή, είναι η στρατηγική η μεικτή. Όλες αυτές οι σκέψεις και πιστεύω ότι θα είχε κανείς πολλά να πει σε αυτό το τομέα και η έκθεση του κυρίου Προύστ δίνει τη δυνατότητα να προετοιμάσουμε πολλές ενδιαφέρουσες απαντήσεις, πολλές προτάσεις βρίσκονται στις τροπολογίες των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκέρεκ. Συνάδελφος Βαλεάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω αυτή την έκθεση, γιατί όντως τονίζει τις ε, ανησυχίε που έχουν αναφερθεί και από την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου που ασχολείται με το θέμα. Νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για την ε, μεταρρύθμιση της ε, προοπτικής για την ευρωπαϊκή πολιτική για την αυτοκίνητο βιομηχανία και πρέπει να καταλήξουμε σε, ένα πλήρες, ε, σε μια πλήρη δέσμη συμπερασμάτων. Ο συνάδελφος στην προσπάθειά του θέλει να προσθέσει συγκεκριμένα εργαλεία και μηχανισμού στην έκθεσή του, αλλά και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την βελτίωση της ευρωπαϊκής αυτοβιομηχανίας. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να ε, στρέψει τις προσπάθειες της Κομισιόν προς το συντονισμό των πολιτικών αντί την στοχοποίηση της ε, ε, αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως θα μιλούμε για το κλίμα, για το εξωτερικό εμπόριο, και εδώ θέλω να πω ότι η Κομισιόν δεν χρειάζεται περισσότερες εξουσίες για να εφαρμόσει τις επιθυμίες της, ούτε χρειάζεται να παράγει περισσότερη νομοθεσία για να κλείσει κάποια κρεμόντα ζητήματα. Η νομοθεσία υπάρχει, τα θέματα είναι γνωστά. Η αυτοκίνητο βιομηχανία και οι καταναλωτές και οι υπάλληλοι χρειάζονται νομική βεβαιότητα, πολιτικό συντονισμό, αλλά δράση πάνω απ' όλα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ότι το σχέδιο δράσης αυτοκίνητα 2020 θα κάνει αυτό που λέει. Η δράση είναι και πάλι το σημείο κλειδί δημιουργώντας μια πλήρως ενιαία αγορά, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, να μειώσουμε την γραφειοκρατία και να δώσουμε αυτή την άμεση δράση που χρειάζεται. Γενικώ πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο και από κοινού να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση και πραγματικά προσβλέπω στην συνεργασία μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Ζαντό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή για την έκθεσή του αυτή. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που κάνει ο εισηγητής, όχι αναγκαστικά με όλα τα συμπεράσματά του βέβαια. Όταν ο εισηγητής μας λέει απόλυτα δικαιολογημένα ότι σήμερα έχουμε μία δυνατότητα υπερπαραγωγής στον τομέα των αυτοκινήτων, δεν νομίζω ότι ε, με τη φράση αυτή δίνουμε τη σωστή απάντηση, γιατί αυτή ε, η κατασκευαστική υπερικανότητα τελικά επηρεάζεται πάρα πολύ από κρατικές επεμβάσεις, δηλαδή από την κρατική υποστήριξη για την τόνωση της ζήτησης. Υπάρχουν πάρα πολλά κρατημέλη τα οποία μέσω bonus, μέσω πριμ, πριμοδοτούν τελικά την ζήτηση των καταναλωτών για αυτοκίνητα, για οχήματα. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση την επιλύει την διαρθρωτική κρίση που πλήττει την αυτοκινητοβιομηχανία. Και τελικά καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη όχι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ένα σημαντικό μέρος των κρατών μελών τελικά βλέπει ότι όλο και περισσότερες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων κλείνουν, ακριβώς επειδή δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Καλείται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πλέον μια συντονισμένη πολιτική εξόδου από την κατάσταση αυτή της υπερβολικής ικανότητας παραγωγής και να καταφέρουμε τελικά να πρικοδοτήσουμε άλλους βιομηχανικούς τομείς με την δυνατότητα αυτή υπερπαραγωγής που υπάρχει στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Να καταφέρουμε δηλαδή, προχωρώντας προς επενδύσεις σε άλλους τομείς, να χρησιμοποιήσουμε άλλους σημαντικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα οι χαλιβουργίες. Να καταφέρουμε να τονώσουμε, αν μη τι άλλο, τις παραγγελίες για άλλους κλάδους, όπως αυτοί οι οποίοι παράγουν συστατικά μέρη των αυτοκινήτων ή ακόμα και για τις εταιρείες εκείνες οι οποίες παράγουν φωτοβολταϊκά Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στρέψουμε επίση περισσότερο την παραγωγή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούμε στους τομείς εκείνους ή σε τα μέσα εκείνα μεταφορά τα οποία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν, να απορροφήσουν ένα μέρο τη δυνατότητα παραγωγή από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν, για παράδειγμα οι Βρυξέλλες ή ε, άλλες πόλεις όπως η Φραγκφούρτη χρησιμοποιούν λεωφορεία με 0% εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά είναι η ε, κινέζικη εταιρεία BYD που παράγει τα λεωφορεία αυτά. Και είναι η ε, δεύτερη σε σειρά εταιρεία η οποία παράγει και τηλεοράσεις ή κάποια άλλα προϊόντα και βλέπουμε ότι τελικά είναι μια κινέζικη εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται να ανταγωνιστεί τις δικές μας εταιρείες. Για ποιο λόγο δική μας η βιομηχανία δεν καταφέρνει να καινοτομήσει προκειμένου να καταλάβει τα τμήματα εκείνα της αγοράς που ανταποκρίνονται ανάγκες που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης για νέα μέσα μεταφοράς για ποιο λόγο να μην καταφέρουμε να κρατήσουμε σε ευρωπαϊκή επικράτεια τόσο τα εργοστάσια και τις μονάδες παραγωγής, όσο και τους υπεργολάβους ή τις υπόλοιπες εταιρείες που παράγουν εξοπλισμό. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο της έκθεσης το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Η διάρθρωση ανάμεσα στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις ρυθμίσεις τις οποίες εμείς εγκρίνουμε τις ρυθμιστικές αρχές. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια διεξάγουμε μία συζήτηση και μάλιστα αποκλίνουν εκεί απόψεις για το αν πραγματικά πρέπει να ρυθμίσουμε τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο στο περιβάλλον που έχουν τα αυτοκίνητα, ιδίως για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό που βλέπω πολύ συχνά είναι ότι τα κράτη-μέλη ακολουθούν τελικά πιστά την στρατηγική την οποία χαράσουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, αποδέχονται ακόμα και τα μεγάλα πολλές φορές ε, δρακόντια μέσα αναδιάρθρωσης τα οποία εφαρμόζουν και βλέπω ότι πολλές φορές ακολουθούμε ιδιαίτερα το παράδειγμα κάποιων μεγάλων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα της ρύθμισης, όσον αφορά το ζήτημα της προστασίας, θα έλεγα το ακόλουθο. Βλέπουμε ότι η διπλωματία της Mercedes τελικά είναι αυτή η οποία κερδίζει. Η εταιρεία αυτή φαίνεται να έχει το πάνω χέρι. Γενικότερα οι γερμανικές εταιρείες. Βλέπω ότι υπάρχουν ε, ιταλικές ή γαλλικές εταιρείες που δεν καταφέρνουν τελικά να επιβάλλουν την άποψή τους στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αυτοκινητοβιομηχανίας και επικρατεί τελικά η άποψη ότι οι δικές τους ανησυχίες δεν εκφράζουν ε, τα γενικότερα συμφέροντα και τις ανησυχίες του ολόκληρου του ευρωπαϊκού κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον για την προστασία του περιβάλλοντος και τουλάχιστον για τους καταναλωτές να καταφέρουμε να έχουμε μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των ε, αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά επίσης και των παράπλευρων συναφών βιομηχανιών. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε έναν ενάρετο κύκλο ανάμεσα στην καινοτομία, τις χαμηλές εκπομπές διοξείδου του άνθρακα και στην ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Συμφωνώ ότι η βιομηχανία είναι μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, σε ένα μεγάλο τμήμα της έκθεσης αυτής αγνοούνται κάποια θέματα που σημαίνει ότι ε, έτσι μειώνεται η ζήτηση ε, ευρωπαϊκώς κατασκευασμένων ε, αυτοκινήτων. Βεβαίως ακόμα βρισκόμαστε στα μέσα της κρίσης, έχει μειωθεί η ζήτηση, είναι λογικό. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι και εμείς φταίμε για αυτή την κατάσταση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε τελικά. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έκανε τελικά για την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας μας. Ρίχνουμε χρήματα στην ανανεώσιμη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυξήσαμε τις τιμές της, ε, της ενέργειας. Η ανταγωνιστικότητα όμως σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις τιμές της ενέργειας. Βγάλαμε τον, από μόνοι μας την Ευρώπη από τις αγορές. οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα επίσης και οι σχετικοί στόχοι που έχουμε θέσει. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Είναι η καλύτερη του κόσμου. Αλλά αυτό έχει και τεράστιο κόστος. Και τα αυτοκίνητα μας έχουν ε, πάρα πολύ ψηλές τιμές ως απόρρια αυτού, γιατί αυτή η τεχνολογία μείωση ε, των ε, εκπομπών διοξιδίου δεν είναι φτηνή. Η δική μου χώρα είναι μεγάλη παραγωγός αυτοκινήτων. Και όταν ε, πηγαίνω στην Τσεχία και μιλώ με τους ε, ε, διευθυντές, με αυτοκινητοβιομηχανίες, με τη Σκόντα για παράδειγμα, μου λένε ότι αν δεν, ήταν, αν δεν υπήρχε η Ασία, η Σκόντα θα βρισκόταν σε ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει λίγο να αναδιπλωθούμε, να ξανακοιτάξουμε την φιλοδοξία που έχουμε, τις φιλοδοξίες που έχουμε θέσει. Εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε νέες τεχνολογίες, είμαι υπέρ του να έχουμε ισχύρια αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τα πράγματα λίγο ψύχρεμα, να δούμε την πραγματικότητα, να σταματήσουμε να βάζουμε το ε, κάρο πριν το άλογο και να σταματήσουμε να επενδύουμε σε ε, ε, τεχνολογίες που ακόμα δεν είναι αποδεδειγμένα υποφελείς. Πρέπει λοιπόν να, να δράσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, κάποιες καταστροφές που στο παρελθόν δεν καταφέραμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ο, Ο Μπερτό τώρα. Άκουσα με προσοχή την ε, ε, εισήγηση. Όντως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και την αμερικανική αγορά. Και θέλω να υπογραμμίσω μια πτυχή σημαντική νομίζω και εκεί μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο η Ευρώπη. Πέρα από την τεχνολογική καινοτομία που σίγουρα η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα ακολουθήσει για ένα σωρό λόγους εμπορικούς, περιβαλλοντικούς κτλ. Θα πρέπει να σταθούμε ε, στην καινοτομία και στην εμπορευματοποίηση των ε, αυτοχήμάτων στο ΣΥΠΑ προωθείται περισσότερο η χρήση του αυτοκινήτου παρά η κατοχή αυτοκινήτου. Και κάνω αυτή τη διαφοροποίηση γιατί σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια γραφειοκρατία γύρω από την κατοχή οχήματος που θεωρείται ως ένα κινητό περιουσιακό στοιχείο καταγεγραμμένο και που καθιστά πολύ δύσκολη την εμπορία αμέσω διόδων πιο ε, γρήγορων. Σκεφτείτε πω αν μπορούσαμε να αγοράζουμε διαφορετικό αυτοκίνητο σε σχέση με αυτό που έχουμε, απλά και μόνο γιατί μέσα στη βδομάδα μπορεί, να χρειάζεσαι ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ενώ στο Σαββατοκύριακο κάποιο άλλο. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται κάποιες ώρες της ημέρας, ενώ ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο κάποιες άλλες ώρες. Θα σκεφτούμε και την εποχικότητα. Λέω η γραφειοκρατία λοιπόν που κινείται γύρω από την κατοχή αυτοκινήτου ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια στρατηγική εμπορική με την ώρα, με το μήνα, με τη βδομάδα ε, και να δημιουργηθεί έτσι μια νέα σχέση ανάμεσα στο χρήση και το αυτοκίνητο που δεν περνά αποκλειστικά και μόνο από την κατοχή ενός ε, αυτοκινήτου που είναι χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής κουλτούρας αλλά από την χρήση του οχήματος που είναι πιο χαρακτηριστικό της αμερικανικής ε, νοοτροπίας. Ευχαριστώ. κύριος Μπέλετ.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 Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προβώ σε κάποιες παρατηρήσεις στα Ολλανδικά. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Συγχαρητήρια στον κύριο Προύστ, Προύστ για την εξαιρετική του αυτή έκθεση. Μπορούμε να δεχτούμε όλα όσα μας παρουσίασε. Όμως θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις επιπλέον όσον αφορά τις ε, ε, την εμπορία που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στρατηγική εναλλακτικών καυσίμων νομίζω πως είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών υποδομών σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν πολλοί που αμφιβάλλουν όσον αφορά το εύρος αυτής της ε, της χρήσης μάλλον αυτής της ε, τεχνολογίας αλλά πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι. Αυτό έχει τεράστια σημασία για την αυτοκινητοβιομηχανία και επίσης μιλάμε για συγκεκριμένα πλαίσια. Ο Επίτροπος Ταγιάννη μίλησε για τον Γαλιλαίο. Ε, ε, υπάρχει και το σύστημα e-call. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα, να μην βαρύνουμε υπερβολικά δηλαδή το σύστημα και να μην πλημμυρίσουμε τον τομέα από ε, γραφειοκρατικά υποχρεώσεις αλλά η σχέση ανάμεσα στο Γαλλαίο και το e είναι εξαιρετική πρωτοβουλία και πρέπει να τη στηρίξουμε. Επίσης η σχέση με τις ευφυείς πόλεις, smart cities. Και αυτή είναι σημαντική. Πρέπει να τονιστεί η καινοτομία. Η καινοτομία όχι μόνο για τις εταιρείε, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα για την αυτοκινητό βιομηχανία. Σημείο 4 τώρα στην έκθεση του κυρίου Προύστα αναφέρεται το συγκεκριμένο στοιχείο είναι το κόστος της ενέργειας για τον κατασκευαστή αυτοκινήτων. Και εδώ συγκρίνουμε την Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια υπέρ των κατασκευαστών αυτοκινήτων της Ευρώπης, γιατί η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή στην Ευρώπη. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν να, δείξουμε, να επιδείξουμε καινοτόμο πνεύμα και να υποβάλουμε προτάσεις που στόχο θα έχουν τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Και να σας πω και κάτι που αφορά την εμπορική πολιτική απέναντι στην Νότια Κορέα για παράδειγμα. Ε, και εδώ ε, ε, θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε διδάγματα και να ε, τα χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο νέων ε, συμφωνιών όπως με την Ιαπωνία να αποφύγουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη και να επιβαρύνουμε υπερβολικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία με υπερβολικά πολλές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλετ. Το λόγο. Ποιος είναι εδώ, εξ ονόματος της Επιτροπής, υπάρχει κάποιος. Κανένας δεν είναι εδώ από την Κομισιόν. Το λόγο έχει λοιπόν ο κύριος Προύστ. Παρακαλώ. Λυπούμε βεβαίω που δεν υπάρχει κανεί εδώ εκπρόσωπο τη Κομισιόν και θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η αντίδραση τη Κομισιόν σε σχέση και σε σχέση με τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων, φυσικά και άκουσα με μεγάλη προσοχή τις διάφορες ε, ε, ποιοτικές παρεμβάσεις. η έκθεση ούτως ή άλλως είναι μια φάση μέσα σε όλη αυτή την πορεία και άκουσα τα όσα είπε ο συνάδελφος Ζαντό για τις διευκρινήσεις που ίσως θα πρέπει να κάνουμε για την νομοθεσία, να επιμείνουμε ας πούμε σε αυτό το τομέα καινοτομία και έρευνα και φυσικά και θα είμαι στη διάθεσή σας έχουμε δουλέψει με το σύνολο των πολιτικών ομάδων για να τελειοποιήσουμε αυτή την έκθεση, να λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες σας, διότι τονίζω και ξανα, τονίζω ότι θέλουμε να δώσουμε ένα αξιόπιστο μήνυμα προς τον έξω κόσμο, θα πρέπει μέσω αυτής της έκθεσης να, να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο και ευχαριστώ τους διάφορους σκιώδει εισηγητές και τους παρεμβαίνοντες σήμερα που εμπλούτησαν αυτή τη συζήτηση και την έκθεση κατά συνέπεια. Ευχαριστούμε κύριε Προύστο. Να θυμίσω ότι η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η Τετάρτη 25 ε, Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και ότι θα έχουμε στη συνέχεια την ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε μια τέτοια μέρα. Ή Είμαστε πολύ γρήγοροι εμείς, είτε πολύ καθυστερημένοι ή, ή προσκεκλημένοι μας. Κάνουμε λεφτά και διάλειμμα περιμένοντας τον Φίλιπ Λόβο που προβλεπόταν στις 11 και 45. πέντε λεφτά διάλειμμα λοιπόν.

Γενικός Διευθυντής της Γενικής ε, Διεύθυνσης Ενέργειας, σχετικά με σχέδια ενεργειακών υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Θα δώσω λοιπόν στον κύριο Λό αμέσως τώρα το λόγο και στη συνέχεια και οι συνάδελφοι εφόσον ε, επιθυμούν μπορούν να πάρουν το λόγο για το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Παρακαλώ. Well, thank you, Chairman. Good. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα στα αξιότιμα μέλη. Ήθελα να σας μιλήσω σήμερα γιατί στις 10 Οκτωβρίου η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια κατεξουδότηση πράξη. Ξέρω ότι ε, ο όρος ε, κατεξουδότηση πράξη για το Κοινοβούλιο είναι σαν το φως για τον ε, ε βρικόλακα, αλλά είναι ένα σημαντικό ορόσημο αυτό για την υιοθέτηση ενός καταλόγου σχεδίων υποδομών κοινού ενδιαφέροντος ότι αφορά την κατασκευή τέτοιων υποδομών στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη και κυρίως ότι αφορά τη διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών. Θα θυμάστε ότι το Κοινοβούλιο έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την ε, διαχείριση των ε, εξελίξεων σε ό,τι αφορά της ανάπτυξης μάλλον των ε, ενεργειακών υποδομών με βάση και την νομοθεσία που δέθηκε σε ισχύ το Μάιο του τρέχοντος. Από κοινού λοιπόν η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν ε, αντικειμενικά κριτήρια και ε, διαφανείς διαδικασίες για να δουν ποια είναι τα σχέδια αυτά που θα πρέπει να λάβουν το καθεστώς ε, σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος. Υπήρχαν βεβαίω και παλαιότερα νομοθετικά κείμενα σε σχέση με το θέμα αυτό, όπου καταλήξαμε τελικά να έχουμε, βάσει των οποίων καταλήξαμε να έχουμε 600 σχέδια που μπορούσαν να θεωρηθούν σχέδια ενεργειακών υποδομών κοινού ενδιαφέροντο, αλλά ουσιαστικά δεν επελέγησαν γιατί ήταν προγράμματα που, ήταν, που είχαν προταθεί από μεμονωμένα κράτη-μέλη και υπήρχε έτσι ε, μια διαδικασία διαιτησίας για να ε, ε, κλέξουμε τα καλύτερα. Καταλήξαμε σε έναν σύντομο κατάλογο, εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το θέμα της κατασκευής υποδομών κοινών ενδιαφέροντος στην Ευρώπη. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε με την συμφωνία πάνω σε 12 διαδρόμους προτεραιότητας. Δεν θα τους αναφέρω όλους, αλλά φαντάζεστε ότι η διασύνδεση βορρά-νότου είναι σημαντικός ε, διάδρομος ε, και στην κεντρική αλλά και στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, η βαλτική ενεργειακή αγορά, οι offshore, πλατφόρμες στη Βόρεια Θάλασσα, τα έξυπνα δίκτυα, η ανάπτυξή τους, η ε, ηλεκτρική διάδρομη επί τη βάση και της ε, ιστορίας που έχουμε, όλες οι διασυνδέσεις ε, αερίου ήταν από την Ανατολή προς τη Δύση και ε, αυτό ήταν πολύ δύσκολο να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Βεβαίω έχουμε το πακέτο τη νομοθετικό για την εσωτερική αγορά και την πρόταση για να μπορέσουμε έτσι να δώσουν μια καλύτερη κατεύθυνση ώστε να έχουμε πιο ολοκληρωμένες αγορές ό,τι αφορά το αέριο. Για την ηλεκτρική ενέργεια ήδη έχουμε 17 ε, από τις 28 ε, αγορές διασυνδεδεμένες. Αυτές όμως οι διασυνδέσεις είναι πολύ σημαντικές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή και βεβαίως να διασφαλίσουμε και τον ανταγωνισμό. Η διαδικασία λοιπόν σύμφωνα με την οποία ο κανονισμός προβλέπει την, τον καθορισμό αυτού του καταλόγου των, των σχεδίων ήταν να, ενός, να συνδέσουμε κάθε ένα από αυτά τα project με έναν από τους διαδρόμους. Και έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι τα σχετικά, τα εν λόγω σχέδια θα είχαν και κάποια ωφέλη τουλάχιστον για δύο κράτη-μέλη. Ότι δηλαδή θα ενισχύουν την συμβατότητα, την ασφαλεία της ε, προμήθειας και θα γίνονταν πάνω σε μια βιώσιμη βάση. Ακόμη και πριν από την επίσημη υιοθέτηση αυτού του κανονισμού ε, και οι περιφερειακές ομάδες και οι εμπλεκόμενοι φορείς άρχισαν να συναντώνται ώστε να επιτεχνηθεί η διαδικασία και να είμαστε ε, σίγουροι ότι ε, στον χρόνο που είχαμε θα, μπορέσου, θα μπορούσαμε μέσα στο 2013 να δημιουργήσουμε αυτόν τον κατάλογο που θα αποτελούσε τη βάση, την κινητήριο δύναμη για να αναπτυχθούν αυτές, αυτά τα σχέδια στην Ευρώπη. Εμείς επικεντρωθήκαμε στον κανονισμό και ε, υιοθετήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο να εξασφαλίσουμε αυτή την άμεση σχέση μεταξύ των σχεδίων και των στρατηγικών συνδέσμων. Δεύτερον, θέλαμε οι εθνικές ρυθμιστικέ αρχές να συμφωνήσουν, να μελετούν σχέδια όχι μόνο ε, σε εθνική βάση για το καλό των ε, δικών του πολιτών, αλλά να έρθουν από κοινού σε ένα τραπέζι και να δουν ποια είναι τα σχέδια που μπορούν όντω να επηρεάσουν μεγαλύτερες περιφέρειες. Δεν είναι κάθε διασύνδεση καλή διασύνδεση, αλλά πολλέ από αυτέ τι διασυνδέσει ήταν εθνικέ λύσεις και αποτελούσαν πολύ πιο ε, ε, δαπανηρή επιλογή από το ότι θα μπορούσε να έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έγιναν λοιπόν διάφορες τέτοιες συναντήσεις μεταξύ ρυθμιτικών αρχών, εμπλεκόμενων φορέων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα κράτη-μέλη ενεπλάκησαν σε αυτές τις περιφερειακές ομάδες έτσι ώστε να καταρτήσουν μια σειρά προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική λίστα, στον τελικό καταλόγο. Ξεκινήσαμε με μια ευρεία διαβούλευση, βασισμένη στην ε, ε, δουλειά των, ε, του δικτύου operators της Ευρώπης. Έγινε μια δημόσια διαβούλευση για το ποια είναι τα projects που μπορεί να είναι χρήσιμα. Ξεκινήσαμε περίπου με 750 τέτοια σχέδια, τα οποία βεβαίως έχουν καταλήξει τώρα να είναι 248 για την ακρίβεια. Αυτός ο κατάλογος των 248 projects θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για να τον εξετάσει στα πλαίσια της διαδικασίας με την της πράξη σε δύο μήνες. Μπορεί να υπάρξει μια παράταση για δύο μήνες ακόμη. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 248 project όπως είπα, αλλά τα project αυτά Ε, καμιά φορά διασυνδέονται μεταξύ τους. Έχουμε δηλαδή περίπου 100, ίσως λίγο πάνω από 100, που αποτελούν κλάστερς, αποτελούν ομάδες. Αλλά πέραν αυτών των 100 που μπορεί να αποτελέσουν ε, ομάδες, υπάρχουν 248 ε, μεμονωμένα σχέδια τα οποία αφορούν κυρίως το αέριο. Η εργασία λοιπόν που έκαναν οι περιφερειακές αυτές ε, ομάδες θα, βοηθήσει ώστε αν αυτά τα σχέδια υιοθετηθούν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επί τη βάση της κατεξόδησης πράξη της ε, Κομισιόν να αποτελέσουν επιλέξιμα project ε, για τον τελικό κατάλογο. Θυμάστε ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε σε 3,5 χρόνια ως νομικό όριο με την βάση της αρχής της ε, νίας τηρίδας, ώστε να μπορέσουν και οι ρυθμιστικές αρχές να ε, ε, συμφωνήσουν για το ποιες θα είναι οι τιμέ που θα επιτρέπονται, να κατανομηθεί, να κατανομηθεί το κόστος, να είναι τα πάντα σαφή και για τις δύο πλευρές. Και τρίτον, αυτά τα project επί της αρχής δίνουν ουσιαστικά το εισιτήριο της χρηματοδότησης έτσι ώστε να υπάρξει η πρόθεση του Connecting Europe Facility. ένα project ε, κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να, τηρεί κάποιες προϋποθε... να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να τύχει χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. αλλά αυτό αντικατοπτρίζεται και στο Connecting Europe Facility. Θα πρέπει να υπάρχει και ενδιαφέρον για, την, ε, ενδιαφέρον για χρηματοδότηση τέτοιου είδους ε, σχεδίων ε, και αυτά συνήθως είναι τα διασυνοριακά σχέδια. Ε, τα σχέδια δηλαδή που η ασφάλεια της, προμήθειας και η εξάλληψη της απομόνωσης είναι σημαντικά στοιχεία. Αυτά λοιπόν τα project είναι πραγματικά ιδιαίτερως ελκυστικά και προσελκύουν βεβαίως και εμπορική χρηματοδότηση. Ο κανονισμός δίνει και στους ιδιώτες επενδυτές μια ασφάλεια για το καθεστώς που θα έχουν αυτά τα σχέδια, καθώς επίσης και το τι διαχείριση θα τύχουν δυνάμει των διαφόρων ε, ρυθμιστικών καθεστώτων, έτσι ώστε να μην υπάρξουν και καθυστερήσεις κτλ. Τώρα, αυτοί οι κατάλογοι θα υπάρχουν πάντα, όχι. Πρέπει να αναθεωρηθούν, ε, αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια. Και σε κάθε περίπτωση, αν ένα project δεν πληρεί και την τελευταία ε, περιβαλλοντική αξιολόγηση ε, ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου, προφανώς εκεί τίθεται θέμα συμφωνίας με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, επομένως θα αποσυρθεί. Έχει γίνει λοιπόν πολλή δουλειά στις περιφερειακές ομάδες ως προς αυτό και σε συνεργασία βεβαίω με τα κράτη-μέλη και τους εμπειρογνωμονές τους. Δεν περιμένουμε λοιπόν ότι από αυτά τα 248 στα επόμενα δύο χρόνια θα καταργηθούν πάνω από 5 ή 6. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποια που είναι λιγότερο όρημα από κάποια άλλα, ας πούμε στη Βαλτική. Υπάρχουν πολύ ε, ανταγωνιστικά μεταξύ τους ε, προγράμματα, τα οποία κυρίως είναι και την παροχή γροπημένου αερίου. Και το μόνο πρόβλημα είναι, είναι τα, τα σχέδια αυτά είναι τόσο καλά που το μόνο πρόβλημα είναι ποιο, θα, ποιο είναι το σημείο που θα ήταν καλύτερο να επιλεγεί. Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Ξέρω ότι έχετε πολύ, δείχνετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον κατάλογο αυτό. Έχουμε έρθει πολλές φορές σε επαφή και σε διμερή επαφή για σχετικά projects. Και βεβαίως περιμένουμε να συνεχιστούν αυτές οι επαφές μαζί σας στα πλαίσια της ολοκλήρωσης αυτού του καταλόγου, ο οποίος θα υιοθετηθεί από την Κομισιόν στις 9 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε Φίλιπ Λόου. Το λόγο τώρα έχει ο συγητής Κορέιρα Ντεκάμπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε Σαρτόρη και ευχαριστώ πολύ Φίλιπ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, θεωρώ πως αυτή η παρουσίαση είναι πάρα πολύ υγιής από δημοκρατικής άποψης και από την άποψη της διαφάνειας και της καθαρότητας των υποθέσεων αυτών. Θα ήθελα να επαναλαμβάνονται και να γίνεται έτσι μια επικοινωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για το πώς προχωράει αυτή η σημαντική διαδικασία. Και επιτός εισηγητής, ε, εγώ δεν είμαι προκατελημένος καθόλου έναντι των ε, κατεξοδότηση πράξεων, ιδιαίτερα σε αυτή την υπόθεση που θα ήταν πραγματικά δυνατόν να μην έχουμε ε, κατεξοδότηση πράξης. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου επιβάλλεται η κατεξοδότηση πράξη. Δεν ε, μας χαροποιούν ιδιαίτερα και γενικά οι ε, κατεξοδότητες συμπράξεις, αλλά εν γέννη είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι ώστε να γνωρίζουμε πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται. Δεύτερον, θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν για την δουλειά που έχει κάνει. Ε, η Κομισιόν ήταν έτοιμη να κάνει αυτή τη δουλειά ε, από τη στιγμή που εγκρίθηκε ο κανονισμός. Ε, υπήρξε η νομική εφαρμογή και τον Μάιο με την, μαζί με την ε, κυρία Σαρτόρη προχωρήσαμε, αλλά η δουλειά όλη αυτή δεν ξεκίνησε τώρα. Είχε ήδη κάνει την εργασία της ε, η ε, Κομισιόν. Ήρθε και είπε ότι στα περιτά και επαναλαμβανόμενα προγράμματα συνδυάστηκαν σε πέντε σύνολα ότι ακόμα υπήρχε επικάλυψη κάποιες φορές και τελικά έχω την αξής ερώτηση να πω. Ξέρετε πως ένα από τα πιο δύσκολα σημεία σε αυτό το κανονισμό, ιδιαίτερα για το Συμβούλιο, ήταν η συμπίεση των προθεσμιών για τη λήψη αποφάσεων ώστε δηλαδή τα κράτη να αποφανθούν για τα διασυνοριακά προσχέδια. Φαντάζομαι πως ακόμα είναι νωρίς για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας που έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εσείς κύριε Γενική Διευθυντά έχετε πληροφορίες για τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για αυτή τη συμπίεση ή είναι ακόμα νωρίς για να έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Grazie, la Ευχαριστούμε. Η κυρία Βάλιαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόου για την παρουσίαση που κάνατε για την ε, διαδικασία επιλογής των σχεδίων ενεργειακών υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Ε, υπάρχουν ανάγκες χρηματοδότησης βέβαια για τα project αυτά και είπατε ότι ε, θέλετε μέχρι το 2014 να ολοκληρώσετε την ιστορική αγορά ενέργειας. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς των σχεδίων αυτών και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Το πρώτο μου λοιπόν ερώτημα έχει να κάνει με τις περιφερειακές ομάδες. Θεωρείτε ότι η αρχιτεκτονική διάρθρωση των περιφερειακών ομάδων διασφαλίζει τελικά την ποιοτική και διαφανή κατάταξη των σχεδίων αυτών σε περιφερειακό επίπεδο ή ότι δίδεται μάλλον μια πολιτική προτεραιότητα και ποιος ήταν ο ρόλος του συμβουλευτικού φορέα που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή. Δεύτερο τώρα ερώτημα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει τα απαραίτητα δεδομένα για το βαθμό ρημότητας των σχεδίων αυτών, καθώς επίσης ε, και το σχετικό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να γίνει ο διασυνοριακός επιμερισμός του κόστους και να, γίνει, και να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάλυσης κόστους-οφέλους, καθώς επίσης και η διαδικασία διοδότησης. Και αν έχετε μια έκθεση προόδου από τους NCOs για την ανάλυση κόστους-οφέλους, τότε θα θέλαμε να έχουμε και τα σχετικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. Κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Λό, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, για την ε, παρουσίαση που κάνετε επίσης. Μα είπατε τι θα γίνει με τα σχέδια αυτά τα οποία δεν συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία καταψήφισε τον κατάλογο των σχεδίων αυτών εξαιτίας ενός συγκεκριμένου σχεδίου το οποίο ήταν ιδιαίτερα αμφίβολο και αναφέρομαι στον τερματικό σταθμό που βρίσκεται πολύ κοντά στην Τεργέστη της Ιταλίας και το σχέδιο αυτό λέγεται ότι μπορεί να έχει πολύ δεινές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Οι περιφερειακές αρχές, καθώς επίσης και οι κάτοικοι της περιοχής, ακόμα και η ίδια η Ιταλική κυβέρνηση, δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί με ακρίβεια όσον αφορά για το σχέδιο αυτό. Νομίζω πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες όσον αφορά το σχέδιο αυτό και για την ένταξή του, την ενσωμάτωσή του στον κατάλογο των εγκεκριμένων σχεδίων. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε σε σχέση με το project αυτό και πώς θα καταφέρετε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις όσον αφορά τον διάδρομο φυσικού αερίου και τον σχετικό κατάλογο PCIs. Έχει επικαιροποιηθεί ο κατάλογος αυτός. Περιλαμβάνεται από τον Αμπούκ, πώς πώ θα επικαιροποιηθεί το κατάλογος PCI. Επίσης, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα τα ποσοστά διασύνδεσης πριν τα σχέδια PCI και μετά τα σχέδια PCI. Δηλαδή, εγώ έχω ασχοληθεί λίγο με το ζήτημα, έκανα μια μικρή ανάλυση και νομίζω ότι δεν ξεπερνάμε το 10% διασύνδεση που ήταν ε, όχι δεσμευτικός αλλά μη τι άλλο κάποιος στόχος ε, στην αρχή του όλου Για μια περιφέρεια όσον αφορά δηλαδή την Ισπανία και την Πορτογαλία, ακόμα και μετά την εφαρμογή των PCIs, θα είμαστε κάτω από το 5%, δηλαδή δεν πετυχαίνουμε καθόλου υψηλή διασυνδεσιμότητα. Τι μπορείτε να πείτε λοιπόν στις χώρες αυτές, η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι χώρες που θα μπορούσαν να εξάγουν ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν επίσης πολύ μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου, ιδίως η Ισπανία. Θα μπορούσαν ε, λοιπόν να διοχετεύσουν την κοινοτική αγορά με τα αποθέματα αυτά. Επίσης, στο όλο αυτό εγχείρημα μιλάμε για hardware και software. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε στη φάση αυτή το hardware, τις υποδομές. Στην έκθεση του κυρίου Κορέα Ντεκάμπος, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε και μια συζήτηση για το software, δηλαδή για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων transmission, μετάδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε και καλύτερα μοντέλα όσον αφορά τις ροές ενέργειας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβίωσε τη συζήτηση στο ζήτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προωθηθεί περισσότερο. Θα μπορούσατε να αναφερθείτε και σε αυτό. Τι κάνουμε δηλαδή για την πτυχή software του εγχειρήματο. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν είναι να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ για το hardware, τότε δεν καταφέρνουμε σπουδαία πράγματα αν δεν ενισχύσουμε και το software, δηλαδή τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των κρατών μελών στην διοχέτευση φυσικού αερίου αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κύριος Σκέλιν, τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Λό για την σαφέστατη παρουσίαση που έκανε. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ε, τα περισσότερα από τα σχέδια αυτά είναι βιώσιμα, σύμφωνα με τον κύριο Λό, και θα πρέπει ε, να δούμε αν τα σχέδια αυτά θα ανταγωνίζονται βέβαια το ένα το άλλο. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, πολύ σωστά ο κύριο Λό αναφέρθηκε σε προγράμματα υγροποιημένου φυσικού αερίου, αναφέρθηκε επίση στην πτυχή τη ασφάλεια του φοδιασμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδίω το να καταφέρουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μα αγωγού σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να μειώσουμε επίση και την εξάρτησή μα από το ρωσικό φυσικό αέριο και να εκμεταλλευτούμε το ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη μείωση, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε σχέση λοιπόν με το LNG, το ευρωπημένο φυσικό αέριο, υπάρχει ένα σχέδιο στη δική μου τη χώρα και υπάρχουν και άλλα σχέδια σε άλλες χώρες βέβαια, ιδίως ε, στα δυτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τα σχέδια αυτά για το ευρωπημένο φυσικό αέριο, τι προτεραιότητα προτίθεστε εσείς να δώσετε, πώς θα προωθήσετε τα σχέδια αυτά σε σχέση και με τους παράγοντες που ανέφερα στην παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπικ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή και να τον παρακαλέσω να μας στείλει και γραπτό στα σχόλιά του αν μπορεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε λεπτομερέστερα να δούμε πώς έχουν δομηθεί όλα αυτά τα σχέδια, όλα αυτά τα projects και Επίσης, πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, αν γίνεται αυτό. Ερώτημα για την Μεσόγειο. Ε, τι γίνεται με τη στρατηγική για τη Μεσόγειο ή με τα χώρες Μαγκρέμπ. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να θέσουμε κάποιους στόχους και επίσης ποια είναι τα project που προλέπονται για αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Grazie, Ο κύριος Κρόλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο λόγο για τις ε, για την παρουσίασή του. Καταρχάς, για την, ε, για την ασφάλεια της ε, προμήθειας. Προφανώς αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την ύπαρξη ή όχι του δικτύου, αλλά το ότι η ενέργεια θα φτάσει στον ε, καταναλωτή. Υπάρχουν ε, διάφορα θέματα όπου σε κάποια ουσίδη υπάρχοντες διασυνδεδεμένους διαδρόμους, ειδικά στο ηλεκτρικό, ε, στην ηλεκτρική ενέργεια, η παροχή υπαρχοντες διασυνδεδεμένου διαδρόμου, ειδικα στο ηλεκτρικο στην ηλεκτρικη ενεργεια η παροχη γινεται προ τη μία κατεύθυνση μόνο και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη για να είναι αμφίδρομη αυτή η παροχή. Αυτό έχει πρόσφατα προκύψει σε σχέση και με το αέριο. Δεύτερον, μιλούμε για, τους εθνικούς, για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που θα πάρουν τον έλεγχο και θα ε, ενδιαφερθούν για το διεθνές ή για το ε, ε, ευρωπαϊκό όφελος αυτό το project. Αυτό όμως υπονομεύει ουσιαστικά τον, το ρόλο που θα πρέπει να έχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο οποίος είναι να ρυθμίζουν την αγορά εθνικά. Ίσως αυτός ο ρόλος να είναι πολύ γενικός ε, ε, που θέλουμε να παίξει ο εθνικός ρυθμιστής. Επίσης, η Κομισιόν έχει κάνει κάποια ανάλυση σχετικά με το όφελος προς τους καταναλωτές άμεσα από την ύπαρξη αυτών των διασυνδεδεμένων διαδρόμων. Και δεν μιλάω μόνο για του μεγάλου χρήστε, για τι βιομηχανίε, αλλά για τα μικρά νοικοκυριά, για το κάθε ένα σπίτι. Τα τελευταία πέντε χρόνια είδαμε ότι λόγω τη οικονομική κρίση ε, το κόστο τη ενέργεια είναι ο τομέα που έχει αλλάξει το, την τάση σε σχέση με την καθημερινή χρήση. Ε, εκεί που τα υπόλοιπα μειώνονται, η χρήση ας πούμε τροφίμων, ε, ειδών ένδυσης κτλ, η ε, ενέργεια αυξάνεται. Υπάρχουν νέα μέτρα, νέες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και λόγω του κόστους η Καταναλωτέ ε, χρησιμοποιούν λιγότερο, όλο και λιγότερο μάλλον, για να προβλέψουν κάτι για το μέλλον. Πρέπει να δούμε επίση τα διδάγματα που έχουμε από τα προηγούμενα projects. Πολλά από αυτά όντως ε, είχαν πραγματικά τεράστια επιτυχία. Αλλά ε, μία από τις βασικές αρχές ό,τι αφορά τα περιφερειακά project είναι ότι τα, αυτά που αφορούν στις ε, απομακρυσμένες περιοχές ε, μπορεί να μην προτιμηθούν λόγω ακριβώς της γεωγραφικής θέσης. Η Ιρλανδία, ας πούμε, είναι στο τέλος ε, ουσιαστικά της, της, του διαδρόμου αυτού διασύνδεσης. Η γεωγραφική λοιπόν θέση ενός, μιας χώρας δεν θα πρέπει να την αποκλείει εκ των πραγμάτων από το να μπορεί να κάνει κάποιες διασυνδέσεις. Ευχαριστώ ο κύριος Μπαλτσίτης. E, σας ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Στην ε, παρουσίασή σας αναφερθήκατε στις βαλτικές χώρες, καθώς επίσης και στον τερματικό σταθμό LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, και είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για την περιοχή μας. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι εμείς εγκρίναμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα σημαντικά δίκτυα ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις και όσον αφορά τον τομέα του φυσικού αερίου βλέπουμε ότι μία από τις προτεραιότητες είναι το πεπιεσμένο φυσικό αέριο. Πώς πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τέτοιων εθνικών σχεδίων. Έχουμε στη Λιθουανία ένα τέτοιο σχέδιο και υπάρχει και ένας τερματικός σταθμός. Το σχέδιο αυτό είναι εθνικό, αλλά πιστεύω ότι έχει μία ευρωπαϊκή πλέον σημασία και εμβέλεια και μπορεί να προωθήσει πάρα πολύ το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρες όπως η Ρωσία. Και βλέπουμε ότι η τελευταία αυτή χώρα έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η Λουθανία πάρα πολύ γρήγορα προχωρά στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού. Εμείς θεωρώ ότι δημιουργούμε αυτή τη στιγμή προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι δημιουργούμε εναλλακτικέ πηγές ενέργειας σε σχέση με τον μοναδικό παροχό μας όλα αυτά τα χρόνια που ήταν η Ρωσία. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους και δίνω πάλι το λόγο στον Φίλιπ Λόου. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στη συζήτηση, διότι πρόκειται για μια ζωντανή και ε, επικοδομητική συζήτηση όλοι συμμετέχουμε. Βλέπουμε την αναπόφευκτη αύξηση των, καυστερών, των τιμών των στερεών καυσίμων λόγω της αυξανόμενης ε, ζήτησης από την Ασία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Ευρώπη ως ε, έναν ε, σταθεροποιητή τιμών κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει και η Ευρώπη να μπορέσει να χειριστεί με τέτοιο τρόπο την ε, κατάσταση ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχουν όλα τα εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις. Ήθελα να πω λοιπόν και τον προτέρων ότι είμαι έτοιμος να επανέλθω μετά από την έγκριση της κατεξοδότησης πράξης για να συζητήσουμε για όλα αυτά, αν αυτό το θεωρείται απαραίτητο. Η δουλειά της Κομισιόν είναι να εξετάσει λεπτομερώς όλα τα κόστη, όλα τα μεμονωμένα project και να εξηγήσουμε τι γίνεται με βάση και τα όσα έχουν ε, μελετήσει ήδη και οι περιφερειακές ομάδες. Έχουν ε, προτείνει, σας είπα από την αρχή, 750 project, τώρα έχουμε φτάσει τα 250 ε, επί τη βάση μιας ε, εξέτασης ακριβώς πάνω σε θέματα όπως ο αντίκτυπος στην τιμή, στον ανταγωνισμό, στην αγορά. Δεν μπορούμε βέβαια να εγγυηθούμε 100% την επιλογή προγραμμάτων που αφορούν την ε, ε, μεταβίβαση, τη διαβίβαση ε, αλλά από την πλευρά του καταναλωτή εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί και θα εφαρμοστούν οι κανόνες. Ήδη υπάρχει δυναμικό σε σχέδια που έχουν ήδη εξεταστεί και με βάση τον αντίκτυπό τους στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις κλπ. Τώρα να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας ε, για την ε, αναφορά που κάνει στην έκθεσή του για το θέμα αυτό, για τον κατάλογο. Δεν ήταν εύκολο να έρθουν με το μέρος μας όλοι οι συμμετέχοντες. οι ρυθμιστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, ναι, έχουν προφανώς εθνικούς στόχους περισσότερο και προσπαθούν να καλύψουν τους εθνικούς καταναλωτές. Αλλά αν κάνουν ανεξάρτητα η μία, η μία από την άλλη τη δουλειά τους, αντί να την κάνουν από κοινού, ε, τότε προφανώς δεν θα ωφεληθούν οι οι πολίτες ε, σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να κάνουν λοιπόν τους, την αξιολόγηση που α πούμε από κοινού. Το να δουλεύει ο καθένας μόνο του στο γραφείο του, στο σπίτι του και στη χώρα του δεν ε, βοηθάει. Ε, υπάρχει πολλή δουλειά που μπορεί να γίνει από κοινού για να προχωρήσουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα projects. Και επίσης τους, βοηθούν και, τους βοηθάει και η υπηρεσία στη Λουβιάνα Έχει σημασία λοιπόν να υποστηρίξουμε τα όσα γίνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά να δώσουμε και την προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής διάστασης. Που όντως θα κάνει τη διαφορά και όντως θα ενισχύσει και τις εθνικές συνθήκες. Ε, εφόσον η ευρωπαϊκή αναγνώριση των εθνικών προτεραιοτήτων για ανάπτυξη ε, υπάρχει, οι χρηματοδοτικές δυνατότητες ε, για εθνικά προγράμματα επίσης υπάρχουν και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου ε, Επενδύσεων. η δουλειά μας μπορεί να γίνει. Βεβαίως εδώ έπρεπε να δούμε γενικότερες επιπτώσεις και στη Βαλτική ας πούμε, για να μιλήσω για αυτό που ρώτησε ο κύριος Μπαλτσίτης. Η Κομισιόν ε, Νομίζω ότι με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων είναι της άποψης ότι ένας μόνος θερματικός σταθμός υγροποιημένου αερίου που θα καλύπτει όλες τις βαλτικές χώρες, αλλά και τις υπόλοιπες γειτονικέ χώρες, όπως Φιλανδία ας πούμε, είναι μια καλή λύση μακροπρόθεσμα. Καλύτερη λύση από το να έχουμε πολλά περισσότερα projects, τα οποία εγγυώνται με την ασφάλεια προμήθεια στις ευρωπαϊκές χώρες σε περιπτώσεις κρίσης, αλλά το θέμα ουσίας είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το θέμα της διακοπής παροχής και να δούμε το πόσο πληρώνει κανείς για αυτή την παροχή. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι ένας μεγάλος θερματικός σταθμός που θα τον μοιράζονται οι χώρες και θα καλύπτει τις βαλτικές αγορές είναι κάτι που θα έχει όντως αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή παροχή και προμήθεια. Γνωρίζουμε βεβαίως και εμείς, όπως και εσείς, ότι υπάρχουν αρκετά καλοί στόχοι στα project που αναφέρατε, αλλά βεβαίως η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική στις βαλτικές χώρες και γι' αυτό έχουμε λάβει τη θέση που έχουμε λάβει σε εθνικό επίπεδο είναι θετικό, αλλά θέλουμε να είμαστε και λίγο πιο φιλόδοξοι και να υπάρξει μια λύση που θα είναι σκόπιμη και για το σύνολο των βαλτικών χωρών. Πάμε τώρα στον εισηγητή σας. Σχετικά με τους operators και την ε, κομισιόν που πρέπει να καταδείξει τα σχέδια που θα κάνουν τη διαφορά, τα διασυνοριακά σχέδια. ζητώντας όχι μόνο από τους operators, επί τη βάση και των δεκαετών αναπτυξιακών σχεδίων τους, αλλά και από το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, έχουμε μια γενική εικόνα του τι μπορεί να γίνει. Και έχουμε και, την, ε, και, την, και τις ενημερώσεις που θα γίνονται Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που είπατε κυρία Βαλεάν για τις πληροφορίες, θα δώσουμε πληροφορίες ε, μαζί με τον κατάλογο που θα θετηθεί με την κατεξοδότηση πράξη για όλα, πληροφορίες για όλα τα project. Σας διαβεβαιώ ότι η, ε, η σειρά που θα λάβει το κάθε ένα ε, δεν είχε βεβαίως να κάνει με καμία πολιτική επιρροή. Με αυτό πάντα προσπαθούμε να το εξασφαλίσουμε. Πρώτα είναι οι promoters, μετά είναι οι operators του συστήματος και μετά έρχεται η άποψη της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής με βάση την οποία κάνουμε την πρότασή μας. Και μετά πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό, και αυτό είναι υποχρέωση μας από τη συνθήκη, τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι αυτό το project μπορεί να προχωρήσει στην επικρατειά τους. Αυτό καταγράφεται και προβλέπεται από την συνθήκη. Παρ' όλα αυτά, δεν είδαμε στο σύνολο της εργασίας που έχει γίνει από τις περιφερειακές ομάδες ένα κράτος μέλος ε, για πολιτικούς λόγους να επιμένει να ε, αφαιρεθεί από τον κατάλογο κάποιο project. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για ένα, πρόγραμμα που ανέφερε, για ένα project που ανέφερε η κυρία Τζόρνταν. Μάλιστα δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος ότι το καταψήφισε το σχετικό κράτος μέλος, γιατί είχε γίνει μια δήλωση για να το, εξασ... διαβεβαιώσουμε αυτού του κράτους μέλους ότι η τελική απόφαση για την τελική, έκθεση της... για την τελική πρόταση της Κομισιόν θα λάβει υπόψη τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ε, του τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου σε ένα άλλο κράτος μέλος. Μπορώ όμως να σας πω ότι επειδή το πρόβλημα, δεν έχει λυθεί, και παρά τις προθεσμίες που είχαμε, δεν θεωρούμε ότι θα, θα απαλληφθούν οι δυσκολίες. Δεν έχουν λυθεί λοιπόν τα προβλήματα, οπότε μάλλον θα πρέπει να κάνουμε μια ε, εξειδικευμένη πρόταση για αυτό το project. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει από κοινού να το δούμε με τους επιτρόπους. Η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 20 Σεπτεμβρίου. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμπεριληφθεί ένα τέτοιο project μέσα σε αυτή την προθεσμία. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά την εταιρεία συμβούλων με την οποία συνεργαστήκαμε, και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τιμήσω υπέρ του δέοντος του συνεργάτες μου, πάντως πραγματικά εμπιστεύομαι περισσότερο τη δική μου ομάδα συνεργατών από ότι την ίδια αυτή την ε, εταιρεία συμβούλων. Γιατί η εταιρεία συμβούλων παρέχει συμβουλές ουσιαστικά δεν γνωρίζουν όλη την τεχνική, όλο το τεχνικό υπόβαθρο και δεν έχουν όλη αυτή την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν οι συνεργάτες μου. Επομένως πρέπει να σας πω ότι την πρόταση την έχει κάνει ο Επίτροπος, εγώ και η ομάδα μου, όχι η Εταιρεία Συμβούλων. Η Εταιρεία Συμβούλων απλώς μας έδωσε κάποιες αναλύσεις, υπέβαλε κάποιες ιδέες, αλλά δεν επευλήθησε καμία περίπτωση δική της απόφαση. Εμείς πάντα επεξεργαζόμαστε τα όσα μας λένε οι εταιρείε συμβούλων, αν σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζουμε αποφάσεις ή προτάσεις τις οποίες τέτοιες εταιρείε υποβάλλουν. Ξέρετε ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δύσκολες, γιατί όπως σας είπα, τις περισσότερες φορές πρέπει να γίνει μία επιλογή ανάμεσα σε ανταγωνιζόμενα σχέδια. Σε άλλες περιπτώσεις ε, δεν έχει ολοκληρωθεί το ίδιο το σχέδιο. Υπολείπονται δηλαδή ακόμα κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι γνωστές και αυτό μας εμποδίζει στο να πάρουμε μια απόφαση. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε εμείς να σας δώσουμε μια κάποια ένδειξη του βαθμού οριμότητας των σχεδίων περιλαμβάνοντας στον κατάλογο. Ωστόσο, αν παραμείνουν στον κατάλογο για μια επαόριστον περίοδο, τότε κάποια στιγμή, αν δεν εφαρμοστούν δηλαδή, θα πρέπει να αποσυρθούν από τον κατάλογο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό λειτουργεί ως δαμόκλειο σπάθη λίγο για τους promoters, δηλαδή ότι αν δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πρότασή τους, τότε κάποια στιγμή θα αποσυρθεί το σχέδιο αυτό από τον κατάλογο. Οι system operators ενισχύουν και αυτοί με τη συμβολή του στην εργασία που λαμβάνει η χώρα και θα πρέπει τα σχέδια αυτά να ενσωματωθούν σε όλες τις εκθέσεις προόδου που θα υποβληθούν όσον αφορά την ανάπτυξη της υποδομής. Και τακτικά θα υποβάλουμε εκθέσεις προόδου, όπως άλλωστε προβλέπεται από την νομοθεσία, από τον κανονισμό. Σε πολλά από τα σχέδια αυτά όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε κάποια στοιχεία τα οποία θα απασχολήσουν σίγουρα πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να σας πω τώρα ότι ε, ο νότιος ε, διάδρομος ε, φυσικού αερίου, το όλο κόνσεπτ αν θέλετε, η αντίληψη γύρω από τον διάδρομο αυτό εξακολουθεί και ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται να πάρει τη μορφή του Ναμπούκο. Έχουμε κάποια σχέδια μικρότερης κλίμακας, αλλά με αρκετά μεγάλη απήχηση. Μία διασύνδεση από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι την, τα σύνορα της Τουρκίας και στη συνέχεια τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ελπίζω ότι μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε μία απόφαση επενδυτική από την εταιρεία, την ΤΑΝΑΠΑ, Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να αρθούν ακόμα όσον αφορά την πρόθεση του σχεδίου αυτού συγκεκριμένα, που όπως σας είπα βασίζεται σε ένα δίκτυο μικρότερων αγωγών από ό,τι είχαμε στον Αμπούκο. Πάντως παρόλα αυτά πρόκειται για μια πρόταση η οποία έχει πλέον εμπορική διάσταση και δεν είναι απλώς θεωρητικός πολιτικός στόχος. Και θα υπάρχει στη συνέχεια μια διασύνδεση από τα τουρκικά σύνορα προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όμως γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια επιλογή των promoters στα πλαίσια ενός κονσόρσιου μιας κοινοπραξίας και η αρχική πρόταση ήταν να περάσει ο αγωγός από την Ελλάδα και την Ιταλία. Αναφέρομαι στον αγωγό TAP, TAP. Βρίσκεται λοιπόν στον κατάλογο των ε, σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και σαφώς θέλουμε να καταφέρουμε να καλύψουμε και χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία που και αυτές περιμένανε ότι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το δυτικό τμήμα του Ναμπούκο που θα μετέφερε φυσικό αέριο μέσω των χωρών αυτών στην Αυστρία και προφανώς θα αποφελούσε και τις χώρες αυτές διέλευσης. Στο κατάλογο μας λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία κυρίως, αλλά και να έχουμε μια δυνατότητα αντίστροφης ροής που να περιλαμβάνει τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, αλλά και την Αυστρία. Οι όροι του παιχνιδιού λοιπόν έχουν αλλάξει όσον αφορά τον λεγόμενο νότιο διάδρομο. Ο νότιος διάδρομος πάντως ζει και βασιλεύει και βέβαια εκφράστηκαν και κάποιες ανησυχίες από τους ε, παραδοσιακούς φορείς παροχής ενέργειας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατανομάζω χώρες, οι οποίες ε, περίμεναν μια διαφορετική εξέλιξη. Αναλύουμε πάντως όλα αυτά τα δεδομένα και στα πλαίσια των εκθέσεων πρόοδου θα είμαστε θέση να σας δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα ανταποκρινόμενος τέλος στα όσα είπε η κυρία Βάλιαν, θα ήθελα να πω ότι ε, πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την κοινοποίηση του καταλόγου αυτού θα δημοσιοποιηθεί και ένα συνοδευτικό έγγραφο, μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήμερα σας υπόσχομαι ότι θα υπάρχει και ένα τεχνικό παράρτημα στο έγγραφο αυτό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ενδεχόμενες επιπλέον πληροφορίες ε, για τις μελέτες κόστους οφέλους, οι οποίες ε, υποστηρίζουν την όλη αυτή προσπάθεια. Τώρα, η διασύνδεση, ο βαθμός διασύνδεσης ανάμεσα στις κεντρικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς έχει ξεπεράσει το 10%. Πήγα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελόνης το 2002 και θυμάμαι πολύ καλά ότι καταγράφαμε τότε τους στόχους αυτούς για την δυνατότητα διασύνδεσης της τάξης του 10%. Το ουσιαστικό πρόβλημα για μας στην Ευρώπη είναι πρώτον ότι πρέπει να συντοπίσουμε ότι η διασύνδεση ήδη υφίσταται πάρα πολύ στο κέντρο της Ευρώπης και πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τα εφιστάμενα δίκτυά μας, αναπτύσσοντας όπως είπα και εσείς όλο και πιο συστήματα και να καταφέρουμε να προσελκύσουμε τους φορείς εκμετάλλευσης σε μία πλατφόρμα και όχι αναγκαστικά σε δύο ή περισσότερες. Και όσον αφορά τώρα τα περιφερειακά προβλήματα, αυτά είναι πιο σημαντικά. Τις ίδιες ανησυχίες με την Ιρλανδία προφανώς έχει και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Θυμάμαι το πρώην πρωθυπουργό σα, όχι ο κύριο Χόης πάντως, όχι ο άμεσος, πρώην, όταν διενύχθη το τούνελ μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θεώρησε ότι ακριβώς για αυτό το λόγο η Ιρλανδία έχει γίνει ακόμα πιο απομακρυσμένη περιφέρεια. Ισχύει πάντως ότι το κέντρο βάρους όλων των επενδύσεων και του εμπορίου βρίσκεται όλο και περισσότερο στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τα απαραίτητα δίκτυα διασύνδεσης για να καταφέρουμε να φτάσουμε και στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες της Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις διασυνδέσεις, για παράδειγμα ανάμεσα στην Βερική Χερσόνησο και την Κεντρική Ευρώπη. Ως προς τη διασύνδεση των δύο αυτών περιοχών έχουμε φτάσει ένα βαθμό διασύνδεσης 6% τουλάχιστον στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά θα μπορούσε ο βαθμός αυτός διασύνδεσης να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό εξαρτάται και από τα σχέδια τα οποία θα υποβληθούν στο μέλλον και από το τι προτείνεται στο πλαίσιο των σχεδίων αυτών. Πάντως υπάρχει σίγουρα η πολιτική βούληση για την αύξηση του βαθμού διασύνδεσης. Τώρα, τα δίκτυα LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική μας ικανότητα όλο και αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουμε την ε, δυνατότητα να κρατάμε πιο χαμηλές τις τιμές φυσικού αερίου μέσω των τερματικών αυτών σταθμών, βλέπουμε ότι η κατανάλωση LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 30% τα τελευταία χρόνια. Και αυτό γιατί η ε, τιμή του σημαντικού φυσικού αερίου, το οποίο προέρχεται από μη ρωσικές πηγές μεσογωγών, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και η κατανάλωση είναι χαμηλότερη λοιπόν διορθώστε με αν κάνω λάθος, εκτός μικροφώνη παρέμβαση, απάντηση, ναι, μα προφανώς ισχύει αυτό που λέτε. Όχι επειδή η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, αλλά η τιμή του άνθρακα πλέον στην Ευρώπη είναι πιο χαμηλή και η τιμή του συμβατικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών δηλαδή έχει μειωθεί και αυτή με τη σειρά τη. Στην πραγματικότητα το φυσικό αέριο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, η επανάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου θα αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στον τομέα της ενέργειας και θα πρέπει πάντως να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την οποία έχουμε πολύ σημαντικές εισαγωγές και χρήση άνθρακα. Προφανώς θέλουμε να δούμε μια αλλαγή στη στάση αυτή και για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε σε ένα πολύ ψηλό βαθμό ακόμα ρηκτά καύσιμα και συγκεκριμένα άνθρακα. Τώρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες υποδομές LNG σε κάποιες χώρες. Ενδεχομένως ναι, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η στάση αυτή. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας θα πρέπει να δούμε όμως και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα σχετικά σχέδια. Πάντως εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι όντως η ανάπτυξη ικανοτήτων και υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να μας βοηθήσει στο να έχουμε μια διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως μέσω του νοτίου διαδρόμου φυσικού αερίου, και μπορεί επίσης να επηρεάσει και την όλη πολιτική που ακολουθούμε όσον αφορά τον άνθρακα. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Προς τον κύριο Ρούμπικ μόνο να απαντήσω ποιες είναι οι βασικές κατευθύνες γραμμές όσον αφορά την Μεσόγειο. Πρώτον λοιπόν, η Κύπρος και οι πιθανές δυνατότητες διασύνδεσης προκειμένου να καταφέρουμε να διοχετεύσουμε μέσω της Κύπρου φυσικό αερίο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι πιο εμπορικά βιώσιμες διασυνδέσεις είναι αυτές με την Τουρκία, αλλά παρουσιάζουν πρόβλημα πολιτικής πλευράς. Υπάρχει πάντως και ένα τίμημα το οποίο πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να καταφέρουμε να εγγυηθούμε την πολιτική αυτή συνεργασία με την Τουρκία, και επίσης πρέπει να δούμε την δυνατότητα χρησιμοποίησης πιθανών κοιτασμάτων αερίου στην Μεσόγειο. Δεν έχουμε κάνει πλήρεις έρευνες για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών και πρέπει να δούμε αν στα δυτικά της Κύπρου υπάρχουν κάποια τέτοια κοιτάσματα τα οποία θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Επίσης η διασύνδεση μέσω την Ισίας, Μάλτας και Σικελίας για την παροχή φυσικού αερίου επίσης πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο, πάντως είναι σημαντική και μακροπρόθεσμα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα για βελτίωση της ενεργειακής μας διασύνδεσης με την Βόρεια Αφρική μέσω της Ιβηρικής Χερσονήσου. Υπάρχουν εκεί πέρα κάποιες καταπληκτικές δυνατότητες για την εισαγωγή και τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα ήταν λογικό πάντως ε, σε μια πρώτη φάση να εστιαστούμε περισσότερο στην Δυτική Μεσόγειο και να καταφέρουμε να, διασυνδέσουμε, να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις μας με την Ιβερική Χερσόνησο, μέσω της Ιβερική μάλλον Χερσονήσου, και να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένως να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, πάντως ελπίζω ότι απάντησα στις περισσότερες. Ευχαριστούμε Φίλιππλο, για τις απαντήσεις σου, τις ε, Εμπεριστατωμένε, Δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικέ για όλου, αλλά πάντω σίγουρα ήταν μακροσκελή η απάντησή σα. Να θυμίσω ότι θα ξανασυνεδριάσουμε στι 3.